And so we start now. Welcome to everybody and a special way to parliamentarians coming from uh, many, many Ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε και ιδιαίτερα καλώς ορίζω τους συναδέλφους από τα εθνικά κοινοβούλια. Ξέρω πως κάποιοι συνάδελφοι έρχονται ακόμα και έχουν αργήσει και η Κομισιόν το ίδιο. Τόσο εμείς είμαστε εδώ πάντως και έχουμε βέβαια και παρουσία του Υπουργού του Λουξεμβούργου της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας οπότε δεν θέλουμε να περιμένουμε έχουμε εδώ τον Κλοντ Μες ε, τον Υπουργό Εκπαίδευσης ε, Νεολαίας ε, και της Εκπαίδευσης προσεχώς ε, έχουμε και την ε, Λουξεμβουργική Προεδρία, βεβαίως. Ε, ήδη έχουν περάσει σχεδόν οι έξι μήνες, κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά και θα ήθελα μετά την εισαγωγή μου να μιλήσω Ιταλικά, έχετε τα ακουστικά και μπορείτε να διαλέξετε τη γλώσσα που θέλετε. Το νούμεράκι που υπάρχει εκεί πέρα, διαλέγετε το κανάλι. και ε, επί τη ευκαιρία ευχαριστήσω και τους Λοιπόν, θα συνεχίσω στα Ιταλικά τώρα. We adopt the agenda. Ε, θα εγκρίνουμε την μισθοδιάταξη. Αυτό αφορά τους συναδέλφους για ε, την Επιτροπή τη δική μας, δηλαδή, του Κοινοβουλίου. Αν δεν υπάρχουν στάσεις, μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο μερικές διατάξεως. Δεύτερο σημείο, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως ό,τι αφορά την διαρμηνία, πως ε, διαθέτουμε όλες τις γλώσσες από και προς. Εντάξει, βρήκατε το κανάλι που αντιστοιχεί στη γλώσσα σας. Έχουμε λοιπόν διερμηνία από και προς όλες τις γλώσσες εκτός από τα μαλτέζικα και τα κροατικά. Όλα τις υπόλοιπες γλώσσες ε, υφίστανται. Μπορούμε να ξεκινήσουμε αναμένοντας τον Επίτροπο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την συνεδρίασή μας από τους αγαπητούς συναδέλφους και φίλου και προσκεκλημένους και του αγαπητούς φίλου του European Youth Forum ότι Είμαστε και εγώ προσωπικά ιδιαίτερα ευτυχής που γίνεται αυτή η πρώτη διάσκεψη διακοινοβουλευτική για θέματα νεότητας και εκπαίδευσης. Ελπίζω πως και την επόμενη χρονιά θα έχουμε μια διακυβερνητική διάσκεψη διακοινοβουλευτική συγγνώμη διάσκεψη πάνω στο θέμα αυτό. Ελπίζω να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στενές σχέσεις ενδιαφέρουσες με τους πιο <clears throat> σημαντικούς εμπλεκόμενους stakeholders αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι βρισκόμαστε τις παραμονές Α, έφτασε και ο Επίτροπος μόλις ξεκινήσαμε παρακαλώ μισό λεπτό να υποδεχτώ τον Επίτροπο Bene. We are... Dear Commissioner, thank you Αγαπητέ Επίτροπο, ευχαριστούμε που ήρθατε στη συνεδρίασή μας. Θα συνεχίσω με τη μητρική μου γλώσσα. Αυτή είναι μια συνεδρία στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας δίχως να στείλουμε μια πρώτη σκέψη στα θύματα των τρομοκρατικών ενεργειών των Παρισίων και να φράσουμε την ελεγγύη μας προς τους Γάλλους αδέλφους. αλλά γνωρίζουμε όλοι πως δεν έχει πληγεί μόνο η Γαλλία αλλά όλη η Ευρώπη. Θα ήθελα να αφιερώσουμε αυτή την συναντρίαση σε πολλούς νέους, σε όλους ειδικά τους νέους που έχασαν τη ζωή τους ε, εκείνο το βράδυ που εκπροσωπούν ε, τα παιδιά που συμμετέχουν στο Εράσμους με τα οποία θέλουμε να ανοίξουμε συζήτηση. Ε, πλήγησαν σε χώρους ε, ε, συνάντησης που ήταν και ε, στόχος των τρομοκράτων. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε το λόγο και να πούμε ότι ανησυχούμε ιδιαίτερα. Θα θυμίσετε την δήλωση των Παρισίων μετά από τα γεγονότα για τον Τσάρλι Εμπρό και ότι υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη και οξυνόμενη φαινόμενος φανατισμός στην Ευρώπη. Υπερθυμίζω μια φράση πολύ στεναρή ότι μετά από την ε, βασική εκτέλεση στο Σάρλ Εμπρό είχαν γράψει ορισμένοι πως ε, τα θύματα ήταν αδελφοί μας αλλά και οι θύτες είναι παιδιά μας Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη και να ξεκινήσουμε ένα διάλογο διαθρησκιακό μεταξύ μας όπως αυτό αναφέρθηκε και στη δήλωση των Παρισίων για να υπενθυμίσω μια φράση αποτελεσματική, ένα πρόγραμμα αποτελεσματικό που το είπε και ο δικός μου πρόεδρος της κυβέρνησης ο Ρέντσι ανήγγειλε ένα πρόγραμμα το οποίο και εφαρμόζει για κάθε ευρώ στην ασφάλεια, ένα ευρώ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το συνολικό πρόγραμμά μας. Έχουμε βάλει του νέου στην επίκεντρο αυτή της πρώτης διακοινωνική μας συνεδρίασης, διότι είναι ζωτική σημασία η στιγμή. Η ανεργία αφορά ένα 25% των νέων στο τελευταίο καιρό στην Ευρώπη. Έχουμε όμω και τα προβλήματα του Νότου και του Νότου Ιταλία, όπου η αυτή το ποσοστό ανέρχεται στο 90%. 3,5 εκατομμύρια είναι αυτοί οι νέοι. Ενώ η εγκατάλειψη των σχολείων αφορά το 11% και περισσότερο από ένα παιδί στα 4 ε, εμπίπτει στο θέμα της κοινωνικής ε, ε το, το, κοινωνικό πέφτει στο πλαίσιο των ε, κοινωνικού αποκλεισμού θεωρούμε ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να έχει μια ευφύ ανάπτυξη, μια ανάπτυξη i4, βιώσιμη, αλλά και η ανάπτυξη, αλλά και η απασχόληση μόνο αν οι νέοι αποκτήσουν εκπαιδευτικά συστήματα ποιότητας, ανώτερης ποιότητας στο πλαίσιο της διαβίου μάθησης αλλά και με δυνατότητα κατάρτισης ε, στο, ε, μετά από το σχολείο πιστώσεις, ε, ε, ε, πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του EQF. γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η πραγματικότητα που εμπλέκει τους νέους που έχουν και πολλές δυνατότητες επιχειρηματικές. Χρειάζεται επίση να δουλέψουμε για πολιτικές κοινωνικής ένταξης, συμμετοχή στην δημοκρατική ζωή. Λαμβάνεις υπόψη είναι αυτές τις εγκάρσεις σχέσεις ε, με όλα αυτά τα θύματα. Αλλά δεν πρέπει να εστιαζόμαστε μόνο σε θέματα απασχόλησης. Χρειάζονται πολιτικές κοινωνικών επενδύσεων στις πρώτες φάσεις της κατάρτισης και στην ποιοτική κατάρτιση. Τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν συμπεριλάβει το θέμα της κοινωνικής ένταξης των νέων στις προτεραιότητες ε, της κυβερνητικές και ορισμένα κράτη. Είναι τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει πολύ σημαντικέ μεταρρυθμίσει τόσο στο πλαίσιο τη εκπαίδευση όσο και τη εργασία. Θα το θέσουν, θίξουν αυτό διάφοροι συνάδελφοι. Ω συνομοθέτη, εμεί οι βουλευτέ, ε, αγωνιστήκαμε για το 40% του προπολισμού του Erasmus, 2, ε, Erasmus Plus για το 2000, 2020, συγκεκριμένε δράσει για το Erasmus Mundus, για τον εθελοντισμό, για πρώτη φορά για τον αθλητισμό και Νομίζω αυτή είναι η άλλη πτυχή, η άλλη πλευρά για το Erasmus Plus. Ε, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτές τις εξελίξεις με την Επιτροπή Απασχόλησης ε, στο πλαίσιο του Horizon 2020 και τα διευθυντικά ταμεία τα οποία έχουν, ε, έχουν δώσει ένα σημαντικό ποσοστό για τους νέους. Θα δούμε, πρέπει να δούμε πώς ε, χορηγούνται αυτά τα χρήματα σε κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποιε εκθέσει πρωτοβουλία, ένα για την πρόθεση τη στρατηγική education and training που παρουσίασε η Κομισιόν και η έκθεση για του νέου 2016-2018. Μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου θα εγκρίνουμε τρει σημαντικέ εκθέσει. Μία για την εκπαίδευση, για τον θρησκευτικό διάλογο, ένα για την επαγγελματική κατάρτιση και τρίτο για την Ευρω... Ε, σχολείο ε, στην Ευρώπη. Ένα έτος λοιπόν εντατικής εργασίας που ξεκινήσαμε για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια, την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και την ε, ψηφιακή, ψηφιακό θεματολόγιο. Το 2016 έχουμε συμπεριλάβει 6 εκατομμύρια επιπλέον για το Erasmus αποκαταστήσαμε τις περικοπές της δημιουργικής Ευρώπης, αλλά θεωρούμε ότι είναι ανεπαρκή ακόμα χρηματοδοτήσεις για την Ευρώπη των πολιτών. Με τις διευθύνσεις ε, εκπαίδευσης θέλουμε να υπάρξει ένα ε, πρόγραμμα για την ηλεκτρονική διδασκαλία και για μια πρωτοβουλία που έχουν προωθήσει οι νέοι μέσω του διαθροτικού διαλόγου, δηλαδή του European Student e-Card. Ελπίζουμε πως ε, σύντομα να εφαρμοστεί αυτή η πρωτοβουλία. Έχουμε το ζήτημα των δεξιοτήτων που, οδήγησε, ε, που ανέφερε η κυρία Τάισεν και υπάρχει και κάτι ακόμα για να ολοκληρώσω. Για μας έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεσμευτήκαμε και στο Στρασβούργο την προηγούμενη Ολομέλεια αυτό της ε, ανθρωπιστικής ανάγκης και της ανθρωπιστικής του φυσικού χαρακτήρα. Το 2016 πετύχαμε το διπλασιασμό των ποσών που δίνονται τόσο για τους πρόσφυγες στα άλλα κράτη όσο και στο πλαίσιο των δράσεων, των δράσεων. Ζητάμε να ανοίξουν διάδρομοι εκπαιδευτικοί τους, για τα παιδιά των προσφύγων στα πανεπιστήμια μας και με τα μαθήματα εξ Περιμένω λοιπόν από τον Επίτροπο μαζί με, τους, με τα όσα πρόκειται να γίνουν για την Ευρώπη 2010 και την διδασκαλία για το 2016. Όλα αυτά ήθελα να σα τα αναφέρω για να γνωρίζετε ποιε είναι οι δραστηριότητέ μα, και να ευχαριστήσω και του προγνώμονε που βρίσκονται ανάμεσά μα, οι οποίοι θα συμβάλλουν σημαντικά σε εργασίε. Όπω ε, είδατε, η διάσκεψή μα δεν μιλάει μόνο για του νέου, αλλά μιλάει με του νέου και το ότι εδώ βρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας του European Youth Forum, Alan Pal, το γεγονό ότι θα μιλήσουμε μετά από του δύο εμπειρογνώμονε από κάθε πάνελ ω πρώτη παρέμβαση πριν από του ελληνικού βουλευτέ και του συναδέλφου μα θα μιλήσει ένα εκπρόσωπο των νέων. Αυτό είναι απόδειξη για το σημασία που δίνουμε στου νέου στην διάσκεψή μα. Όσοι θέλουν να παρέμβουν, θέλουν να συμπληρώσουν ένα έντυπο το οποίο έχουν μπροστά τους, στο έδρανό τους, αναφέροντας ε, σε ποιο πάνελ θέλουν να παρεύουν. Μετά το τέλος κάθε πάνελ θα διεξαχθεί συζήτηση και θα δώσω στο λόγο ανάλογα με το χρόνο που θα έχουμε διαθεσή μας. Ο πρώτος θα λάβει το λόγο, είναι ένας νέος. Στις 12.30 θα πρέπει να διακόψουμε και θα κάνουμε και μια family photo, μια οικογενική φωτογραφία όσους ήθιστε και μετά θα υπάρξει ένα γεύμα. Θα δώσω αυτή αμέσω το λόγο, Ευχαριστώ τον Κλοντ Μάσου, ε, Υπουργό Εκπαίδευση και πολλών άλλων ζητημάτων. Έχει πολλέ αρμοδιότητε από τη Λουξεμβουργική κυβέρνηση. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, εθνικοί και ευρωβουλευτές. Τι θέση δίνουμε στους νέους στην Ευρώπη σήμερα. Πώς δημιουργούμε για αυτούς τις καλύτερες συνθήκες έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να συνεισφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι βασικά ερωτήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη. Είναι επίσης ερωτήσεις στις οποίες θελήσαμε κατά τη διάρκεια της Λουξιβοϊνής προεδρίας να δώσουμε απαντήσεις μέσω ε, εκθέσεων, ευρωπαϊκών εκθέσεων στον τομέα της ε, ε, νεότητας και της εκπαίδευσης και επίσης με την υιοθέτηση ενός προγράμματος εργασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την νεότητα. Η κατάσταση των νέων στην Ευρώπη είναι τόσο διαφορετική ε, μεταξύ των χωρών όσο διαφορετική είναι και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ορισμένα ζητήματα είναι θεμελιώδη. Μεταξύ αυτών η υπηκότητα, η ευρωπαϊκή υπηκότητα. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε οι νέοι να μπορούν να αναπτύσσουν τις προοπτικές τους και να έχουν μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις μέσω διαλόγου με τους νέους και υιοθετώντα ένα ψήφισμα για την πολιτική συμμετοχή των νέων. Για να ενισχύσουμε την υπηκότητα μέσω της συμμετοχής είναι καταρχήν απαραίτητο να βελτιώσουμε ουσιαστικά τις ε, απόψεις ε, ε, των, αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις σε ό,τι αφορά τους νέους και τη συμμετοχή τους. Θέλουμε όμως να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε και την εκπαίδευση για την ε, υπηκότητα στην Ευρώπη. Έχουν αναλυθεί πολλές πρωτοβουλίες αλλά θα πρέπει να συστηματοποιηθούν και να συντονιστούν. Να ενισχύσουμε τις εταιρικέ σχέσεις ε, μεταξύ της επίσημης εκπαίδευσης και της μη άτυπης εκπαίδευσης είναι προτεραιότητα στο σχολείο αλλά και αλλού ε, θα πρέπει ε, η νεότητα να παίξει σημαντικό ρόλο. Να ενισχύσουμε την επικότητα η ενίσχυση της επικότητας θα πρέπει να ωφελήσει όλους τους νέους. αυτό αποτελεί πρόκληση γιατί οι Ευρωπαίοι νέοι εποφελούνται σε μεγάλο βαθμό των συστημάτων εκπαίδευσής τους αλλά όχι όλοι. Γνωρίζουμε ότι τα εκπαιδευτικά μας συστήματα μπορεί να, είναι, να εντάσσουν περισσότερο τους νέους, να τους συμπεριλαμβάνουν περισσότερους νέους ε, και αυτούς που έχουν προέλθει από τη μετανάστευση. Γι' αυτό το λόγο οι Υπουργοί Εκπαίδευσης ε, ε αποφάσισαν να δράσουν πιο αποφασιστικά ε, σε ό,τι αφορά το θέμα της σχολικής εγκατάλειψης. Η πρόκληση είναι μεγάλη. Αν είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να ε, αντιμετωπίσουμε προβλήματα ριζοσπαστικοποίησης ορισμένων κομματιών της νεότητας ε, ε, είναι επίσης αυτό οφείλεται στο ότι πρέπει να δώσουμε ταυτόχρονα προοπτικές σε όλους τους νέους. Ορισμένοι έχουν την εντύπωση ότι οι ιδεολογίες, ακραίες ιδεολογίες στους αντίποδες των δικών μας αξιών δίνουν περισσότερες απαντήσεις από ότι εμείς. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί. Οπότε η προτεραιότητα του, προ... προτεραιότητες του προγράμματος Εργασία για την νεότητα για τα επόμενα τρία χρόνια είναι η κοινωνική ένταξη των νέων, η συμμετοχή τους και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Αυτές οι τρεις ως τρεις δέσμες ενός κοινού προγράμματος. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασία, ορισμένοι δείκτε ε, φαίνεται ότι δείχνουν ότι ε, έχουμε κάνει ένα βήμα, σημαντικό βήμα, σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων ιδιαίτερως. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε Προ την ίδια κατεύθυνση και αποφασιστικά. Με το σχήμα, με, το, με την εγγύηση για την νεότητα, ε, δώσαμε στον εαυτό μας ένα σημαντικό εργαλείο για να συντονίσουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες στον τομέα της εκπαίδευση της νεότητας και της απασχόλησης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την εφαρμογή αυτού του συστήματος. Θέλω όμω να σα μιλήσω και για την κατάσταση των μεταναστών στην Ευρώπη, ιδιαίτερω αυτών που έχουν φτάσει πρόσφατα το 2015 ήταν δραματική χρονιά. Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα συνέρευσαν και συνεχίζουν να σειραίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δημιουργεί προβλήματα που πρώτη φορά βλέπουμε, μεταξύ άλλων στα εκπαιδευτικά συστήματα. Πώς μπορούμε να στηρίξουμε την ένταξη όλων αυτών των νέων μεταναστών, οποιαδήποτε και αν είναι η διάρκεια ε, διαμονής του στην Ευρώπη. Αποφασίσαμε εντάχει να αφιερώσουμε το, τις του επόμενου ε, Συμβουλίου Υπουργών ε, Νεότητας Εκπαίδευσης ε, Πολιτισμού και Αθλημάτων σε αυτό το θέμα. οι συζητήσεις έχουν δείξει ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τους μετανάστες μέσω των εκπαιδευτικών συστημάτων, να προωθήσουμε τον διαπολιτισμικό διάλογο, να ενισχύσουμε την δημοκρατική συμμετοχή και ιδιαίτερως να βοηθήσουμε τους πιο αδύναμους για να συνεισφέρουμε με τους συναδέλφους του Συμβουλίου ε, ε, του Λεξεμβούργιου συναδέλφους του Συμβουλίου έστειλα ε, στους πρόεδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τι, τα συμπεράσματά μας ελπίζοντας ότι θα αναλυθεί η δράση. Κυρίε και κύριοι αυτά εισαγωγικά ε, μια επισκόψη των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε και θα πρέπει να λύσουμε. Καλή επιτυχία και ένα καλό διάλογο. Thank you so much for your Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και την δέσμευση αυτή που αναφέρατε. Φαντάζομαι πως θα αποτελέσει θέμα της συζήτησης για τις συγκεκριμένες αυτές δεσμεύσεις επειδή πρέπει να προλάβουμε την ριζοσπαστικοποίηση και τον αποκλεισμό Μιλήσαμε και στην προηγούμενη Ολομέλεια για μια κοινή προσέγγιση στην Ευρώπη έτσι ώστε τα αγόρια και τα κορίτσια αυτά να έχουν κάποια στήριξη. Γι' αυτό και κονδύλια. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε για αυτή τη δέσμευση. Τώρα δίνω τον λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Ναύρατσιτς. Γνωρίζετε πως είναι Επίτροπος ε, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, ε, Νεολαίας και Αθλητισμού. Λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες ε, σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφερθώ στον ρόλο της εκπαίδευσης και της πολιτικής για την νεολαία για να αντιμετωπιστεί η ριζοσπαστικοποίηση και ο αποκλεισμός ε, των ε, νέων. Οι κτηνώδεις αυτές επιθέσεις ε, που έγιναν στο Παρίσι μας υπενθυμίζουν τις ε, εντάσεις ε, στην κοινωνία μας που εκτιλήσονται σε μία ήπειρο που ακόμα αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο κοινωνικός ιστός διαλύεται. Πάνω από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και η ανεργία των νέων ακόμα απαράδεκτα υψηλή. Η ένωση μας ε, τώρα είναι λιγότερο ίση. Βλέπουμε ένα χάσμα. Για πολλούς νέους είναι δύσκολο να φανταστούν και ένα λαμπρό μέλλον. Ναι, συνολικά αυτή η νέα γενιά είναι πιο εκπαιδευμένη και διασυνδεδεμένη από οποιαδήποτε άλλη πριν από αυτήν. Πολλοί νέοι όμως θεωρούν ότι ακριβώς τη στιγμή που θέλουν ε, να σταθούν στα πόδια τους, οι ανάγκες τους ε, και οι ελπίδες τους ε, αγνοούνται. Και εγώ συμπάσχω με αυτούς που θεωρούν ότι δεν έχουν ευκαιρίες και Βεβαίω ε, τα όνειρά τους ε, παραμελούνται. Βλέπουμε πως οι νέοι απομακρύνονται από την παραδοσιακή δημοκρατία. Π.χ. πέρσι στις, ε, στις τελευταίες ένα στους τρεις νέους μόνο ψήφισε. Και ακόμη πιο ανησυχητικό, οι νέοι γεννούν την πλάτη τους στις αστικές και δημοκρατικές αξίες, στι οικογένειες και στους φίλους τους. Και έτσι πλησιάζουν πιο κοντά στη ριζοσπαστικοποίηση και την βία εγώ όμως δεν θα δεχτώ να χάσουμε αυτούς τους νέους. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτούς ε, τα επόμενα χρόνια και όχι να περιμένουμε την επόμενη τρομοκρατική επίθεση. Πρέπει να συνεργαστούμε μαζί για την αλλαγή. Εγώ θέλω σε μια Ευρώπη όπου όλοι θα βρουν την θέση τους και θα ζούμε σε ανοιχτές ε, κοινωνίες με ένταξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οικοδομηθεί σε κάποιες ε, θεμελιώδεις αξίες από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σεβασμός της αξιοπρέπειας, ελευθερία έκφρασης, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αξίες αυτές απειλούνται, όπως έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα, και πρέπει όλοι να δράσουμε στο τοπικό επίπεδο, στις κοινότητες, στο περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο οι τομείς ε, αρμοδιότητάς μου, εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στην κοινωνική ένταξη καθώς επίσης και στην πρόληψη της διακριτικής μεταχείρισης. Την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συνάντηση με τους υπουργούς επαναβεβαίωσα τη διάθεσή μας να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. και τα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Είπα πως πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο την κοινωνική ένταξη στους τομείς αρμοδιότητάς μου. Με τους Υπουργούς ε, Παιδείας συμφώνησα σε νέες προτεραιότητες ε, για την εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων την συμμετοχική εκπαίδευση. Οι Υπουργοί Νεολαία συμφώνησαν στο να εστιάσουμε στους νέους την κοινωνική ένταξη όλων και Βεβαίω ε, θα πρέπει οι νέοι να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο στη δημοκρατική ζωή και να μπορούν να περάσουν ευκολότερα στον κόσμο της εργασίας. Όσον αφορά την εκπαίδευση, πρέπει να δούμε το τι διδάσκεται στα σχολεία μας. Οι νέοι πρέπει να έχουν τις δεξιότητες που απαιτείται για να βρουν δουλειά. Η απασχόληση εξακολουθεί να είναι η καλύτερη αντιμετώπιση του αποκλεισμού. Όμως πρέπει να κάνει και περισσότερα εκπαίδευση. Πρέπει να βοηθήσει τους νέους να ασπαστούν τις δημοκρατικές αξίες. Πρέπει να προωθήσουμε τον διαπολιτισμικό διάλογο και κανένα να μην μένει πίσω λόγω πολιτισμικού ή θρησκευτικού ή κοινωνικού υποβάθρου. Και πρέπει να βοηθήσουμε τους δασκάλους. Έχουν πολύ δύσκολες δουλειέ και αντιλαμβάνονται ίσως τους νέους περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν στις δύσκολες συζητήσεις που γίνονται στην τάξη, να αντιμετωπίσουν ακαθόδη ζητήματα όπως τις διαφορές των πολιτισμών, τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση. Γι' αυτό οι δάσκαλοι χρειάζονται πολύ καλή κατάρτιση στον τομέα της νεολαίας. Πρέπει να φροντίσουμε οι νέοι από διαφορετικούς πολιτισμούς να μπορούν να έχουν διαπολιτισμικές επαφές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Από τις δικές μου εμπειρίες γνωρίζω τι μεγάλη σημασία έχουν οι προσωπικές σχέσεις για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και ακριβώς οι εθελοντές και τα πρότυπα σε τοπικό επίπεδο παίζουν εδώ πέρα σημαντικό ρόλο οι φίλοι, οι, οι εθελοντές, οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι στον τομέα της θρησκείας κτλ. Πρέπει λοιπόν να βοηθηθούν όλοι αυτοί. Το 2016 το πρόγραμμα Erasmus Plus θα δώσει περισσότερη χρηματοδότηση σε έργα κοινωνικής ένταξης μέσω της εκπαίδευσης, κατάρτισης, ε, νεολαίας και αθλητισμού. Γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε σε διεθνή προγράμματα και συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων νεολαίας αθλητισμού και πολιτισμού με ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία. Επίσης ε, φροντίζω το πρόγραμμα Erasmus Plus να οδηγεί σε περισσότερη κινητικότητα δασκάλων, ανταλλαγές νέων και διεθνείς συνεργασίες. Τα έργα τα οποία στηρίζουμε δείχνουν ήδη τι είναι δυνατόν. Χρηματοδοτούμε έργα που παραδείγματος χάρη συνδυάζουν την άτυπη εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την κατάρτιση έτσι ώστε την Ευρωπαίοι οι οποίοι δεν δουλεύουν ή δεν εκπαιδεύονται να είναι πιο απασχολήσιμοι. Προσπαθούμε έτσι να ενδυναμώσουμε την νεολαία για να αποφευθεί η ριζοσπαστικοποίηση. Έργα όπως αυτά χρειαζόμαστε και θα στηρίξουμε. Πριν ε, τελειώσω να πω δύο λόγια για το πώς ε, η πολιτική της εκπαίδευσης μπορεί να, ενσωματώ, να βοηθήσει την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών και πράγματι πρέπει να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα για να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικώ. Πέρα από την επίσημη εκπαίδευση πρέπει να μπορούν να εποφελθούν από δραστηριότητες όπως ο εθελοντισμός αλλά και ο μαζικός αθλητισμός. Στηρίζουμε τα κράτη-μέλη σε αυτό. Παραδείγματος χάρη, βοηθούμε τους μαθητές να μπορούν να καταγράψουν τα προσόντα τους στο συντομότερο δυνατόν. Γι' αυτό και φιλοξενήσαμε μια συνάντηση των Εθνικών Κέντρων Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων. Μοιράστηκαν τι υπηρεσίε τους όσον αφορά την αναγνώριση των πτυχίων των προσφύγων. Επιπλέον, αυτά τα οποία τα μαθήματα τα οποία βρίσκονται στο διαδίκτυο στο Erasmus Plus είναι προσβάσιμα από τους ε, πρόσφυγες ε, και τους ε, μεταναστές. Όλοι λοιπόν έχουν να συνεισφέρουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα, τοπικές και περιφερειακές αρχές, κοινωνική εταίροι και κοινωνία των πολιτών. Το κύριο βάρος αυτής της προσπάθειας θα γίνει στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και στα κέντρα νεότητας στις κοινότητές μας. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να εφαρμοστούν τα σχέδιά μας. Αλλά πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Όπως οι δυνάμεις ασφαλείας ε, συνεργάζονται για να κατανικήσουν τους τρομοκράτες, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τα πολιτικά κέντρα και με τους αθλητικούς συλλόγους για να καταπολεμήσουν τον αποκλεισμό, τη φτώχεια και την ανεργία. Κοινωνική ένταξη πρέπει να είναι η απάντησή μας εάν θέλουμε μια Ευρώπη με συνοχή με ανταγωνιστικότητα και σας χρειαζόμαστε και βασίζομαι στην στήριξή σας. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ σοβαρή η δέσμευσή σας. Ξέρετε ότι συμφωνούμε. Ίσως θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερο στένος. Παραδείγματος χάρη στο Erasmus Mundus εμείς ε, δίνουμε προτεραιότητα τα προγράμματα που για τα παιδιά που από αυτές τις χώρες ε, παραδείγματος χάρη περισσότεροι πόροι για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ε, στέσαμε στον προπολισμό αλλά λυπούμεθα που για την Ευρώπη των πολιτών δεν μπορέσαμε να πάρουμε περισσότερα και φυσικά αυτά είναι θέματα πολύ σημαντικά όπως και η ασφάλεια βασίζομαι σε μια συμμαχία με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά θα πρέπει και η Κομισιό να είναι πολύ πιο αποφασιστική και να δεσμευτεί περισσότερο, διότι κάπως μας ανησυχεί το θέμα. Να δώσω το λόγο τώρα στο Γενικό Γραμματέα του του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας Αναμπόλ αλλά πρέπει να υπενθυμίσω ότι οι Φιλανδοί συνάδελφοι που για λόγους υγείας δεν μπορούν σήμερα να διασφαλίσουν την συνέχιση της διερμηνίας στην γλώσσα αυτή, στα φιλανδικά δηλαδή. Παρακαλώ, επόμενος αγορτής έχει το λόγο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συμπληρώστε το έντυπο προκειμένου να μας δηλώσετε σε ποιο πάνελ θέλετε να συμμετάσχετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, Επίτροπε, Υπουργέ. Συχνά λέγεται ότι είμαστε η πρώτη γενιά στην ιστορία ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα πιο δύσκολα. Όντως ε, οι νέοι και τα παιδιά κινδυνεύουν να γνωρίσουν την ε, περιθωριοποίηση. Ε, βρισκόμαστε το 2015 και ακόμα μιλάμε για οικονομική και δημοσιονομική κρίση διότι δεν έχει λήξει ακόμα. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους από το πάνελ που θα στήριξουν διάφορες Δεν θέλω να σας υπενθυμίσω μια ακόμη φορά ότι τα πράγματα είναι άσχημα για τους νέους. Ζούμε σε περίοδο κρίσης και η πολιτική αντιμετωπίζει προβλήματα. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν προβλήματα τα οποία μπορούν να επιληθούν εύκολα και γρήγορα. Τα πράγματα λοιπόν είναι ιδιαίτερα ε, σκοτεινά για τους νέους από οποτεδήποτε άλλοτε στον παρελθόν. Η Ευρώπη υφίσταται πιέση και το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε σε αυτό πως μας είναι αν, χρησιμοποιούμε, αν δημιουργούμε μια Ευρώπη αδύναμη ή μια, μια Ευρώπη ανθεκτική συγγνώμη ή μια Ευρώπη της παραφωνίας. Στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων δυστυχώς δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας ε, την ε, δυνάμεις και των νέων και των μελλοντικών γενεών θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές για τους νέους που θα βασίζουν σε τρία βασικά κριτήρια. Θα πρέπει να είναι ε, ε, εγκάρσιες και συμμετοχικές. Αυτά θα δώσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων. Το, ε, το φόρουμ μας, οποίο συμμετέχουν πάνω από 100 ε, νεολαίες προσπαθούν ε, να δημιουργηθεί μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις όπως τρομοκρατία, ριζοσπαστικοποίηση, μετανάστευση ακόμα και οι ελευθερίες όπως αυτή της ελεύθερης γνώμης και της ελεύθερης έκφρασης. διαρωτώμε. όμως αν θα πρέπει να εκπλαγούμε για την κρίση αυτή που μας πλήττει δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναμένουμε ακριβώς διότι υπήρξε έλλειψη επενδύσεων για τους νέους και τώρα είναι η ώρα για να γίνουν επενδύσεις που αφορούν στους νέους, τους νέους εργαζόμενους και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να πετύχουμε μεγαλύτερη στήριξη αυτών των οργανώσεων που σχετίζονται με τους νέους. Η εκπαίδευση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο ολιστικό τόσο στο άτυπη μορφή εκπαίδευσης για να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις δύο από τους τρεις οργανώσεις των νέων αντιμετωπίζουν προβλήματα με το θέμα της κοινωνικής, ε, Το κοινωνικό πολιτισμού. Τώρα αναφέρεται ότι θα πρέπει οι νέοι να αποκτήσουν δεξιότητες ε, αντίστοιχες με τις ανάγκες ε, της αγοράς εργασίας. Επίσης, ε, όταν μιλάμε για εκπαίδευση, τα... συχνά αυτή γίνεται με τρόπο ακατάλληλο και δεν μπορούμε να περιμένουμε επιτυχία τη στιγμή που υπάρχουν ε, προβλήματα σε μία από τις τρεις ε, οργανώσεις των νέων. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε από όλα τα επίπεδα των εμπλεκομένων να φροντίσουν να υπάρξει κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων. Πιστεύω ότι οι νέοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ στο να συμμετάσχουν στην λήψη αποφάσεων. Δεν αρκεί να πηγαίνουν να ψηφίζουν κάθε φορά που προκυρήσονται εκλογέ. Δεν θα πρέπει λοιπόν να τους παραβλέπουμε τους νέους. Ελπίζω να επαναληφθούν τέτοιες συνεδριάσεις και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Uh, thank you so much. I appreciate your... Ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας. Χρειαζόμαστε, χρειάζεται λοιπόν ε, να σκεφτούμε τις προτάσεις σας. Θα τις συζητήσουμε φυσικά και τώρα. Ε, να πω ότι έχουμε 15 λεπτά Προς το παρόν κανένα μέλος από το Εθνικό Κοινοβούλιο δεν, έχουν, δεν έχει ζητήσει το λόγο. Διότι έχει σημασία να γίνει αυτή η συζήτηση. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ανάμεσά μας τον Υπουργό και τον Πίτροπο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, οι εθνικοί βουλευτές και μετά οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές. κάντε ένα νεύμα που θέλετε να μιλήσετε και έτσι να μπορέσουμε να γράψουμε τα ονόματά σας, να σας καταγράψουμε. Πρέπει να συμπληρώσετε το κίτρινο χαρτί που έχετε μπροστά σας για Ντουσέ από τη Γαλλία. Άλλοι. Άλλος. κυρία Φεράιαν, Νάικοφ, ο κ. Γραμματικάκης για το πρώτο πάνελ και μετά έχουμε τα υπόλοιπα. Η κυρία Ντουσέ έχει το λόγο, παρακαλώ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, ιδιαίτερα για τα λόγια σας και τις σκέψεις σας για τους ε, Γάλλους ε, νέους και αλλά και για την Ευρώπη γενικότερα που ε, εξεπλάγησαν, συνταράχθηκαν από τα γεγονότα του, της 13ης Νοεμβρίου στο Παρίσι και ο συναδελφός μου, Yves Ιβ ε, που είναι επίσης παρόν εδώ δίπλα, ε, σας ευχαριστεί εξίσου. Σε ό,τι αφορά την νεότητα, το θέμα της ε, νεότητας ε, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σήμερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που διοργανώσατε αυτή τη συνάντηση. Θα ήθελα να μιλήσω για το Erasmus Plus. Με την ε, διεύρυνση των δυνατοτήτων κινητικότητας που δίνει. Θέλω να υποστηρίξω αυτή την ιδέα ε, και την, τον εκδημοκρατισμό του συστήματος κινητικότητας, του συστήματος Εράσμους. Ε, λειτουργεί καλά και για το πανεπιστημιακό τομέα και για τους φοιτητές και για το προσωπικό ε, και θα πρέπει να διευρυνθεί και σε άλλους τύπους κοινού, πιο νέους, για παράδειγμα αυτούς τους νέους που βρίσκονται σε μαθητεία, ε, τους νέους των τεχνικών γυμνασίων και λυκείων, τους νέους ε, της ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 500.000 νέους που είναι εκτός εκπαίδευσης και εκτός, ε, και κατάρτισης και έχουμε και ε, ένα παράλληλο σύστημα της εγγύησης για την νεολαία που αρχίζει να λειτουργεί. Θα πρέπει η κινητικότητα να αποτελεί ε, ένα μέσο όχι μόνο για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής συνείδησης αλλά και για να δείξουμε στους νέους ένα ευρωπαϊκό δρόμο προς την απασχόληση. Πρόεδρος, οι απαντήσεις στο τέλος. Δίνω το λόγο στον επόμενο μιλτή. Σαμπίν Φράιαν. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ που έχουμε σήμερα αυτή την δυνατότητα για μια ανταλλαγή απόψεων με τους εθνικούς συναδέλφους για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε εντατικά γιατί ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης έχουμε περιορισμένες αρμοδιότητες ως Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή των περισσότερων πρωτοβουλειών είναι εθνική. Παρ' όλα αυτά, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Ένωση Έχουμε κάποια σημαντικά στοιχεία που πρέπει να δούμε, όπως αναφέρθηκαν, π.χ. τα προγράμματα Erasmus, το πρόγραμμα Erasmus Plus, τα υποπρογράμματα Κομένιους και Leonardo da τα οποία προωθούν τις ε, διεθνείς ανταλλαγές ε, στον τομέα της εκπαίδευσης. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που ε, αναφέρθηκε και θα ήθελα να ρωτήσω ήταν το ζήτημα της ένταξης ε, ανθρώπων ε, μεταναστών. Όχι μόνο των προσφύγων αλλά και αυτών που ζουν χρόνια στις ε, χώρες μας γιατί τα προβλήματα έχουν εκδηλωθεί εδώ και καιρό. Οπότε το ζήτημα είναι με ποια μέτρα θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι όταν έχουμε περιορισμένα κονδύλια Πρέπει λοιπόν με τα εθνικά προγράμματα και εθνικές ε, πρωτοβουλίες να φροντίσουμε αυτό, για αυτό το θέμα. Και αυτό δεν αφορά μόνο την επίσημη εκπαίδευση, αλλά και την άτυπη, όπως αναφέρθηκε και από κάποιον εκπρόσωπο της νεολαίας. Και βεβαίως πρέπει να δούμε τα προγράμματα αυτά. Βεβαίως το ε, κλασικό παράδειγμα είναι το Εράσμος που αφορά την επίσημη εκπαίδευση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την άτυπη εκπαίδευση στο μέλλον. Πολλά από τα προβλήματα της ριζοσπαστικοποίησης δεν είναι ζήτημα επίσημης ε, εκπαίδευσης ή έλλειψης αυτής. Έχουμε νέους οι οποίοι έχουν πολύ καλό ε, και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης αλλά είναι και θέμα έλλειψης ε, προοπτικών. Ε. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Είναι νέοι οι οποίοι θεωρούν ότι δεν έχουν παραδείγματο χάρη ε, επαγγελματικές προοπτικές, αλλά το θέμα είναι η μετάδοση των αξιών που είναι ελληματική στο σχολείο. Το ερώτημά μου λοιπόν προς εσάς είναι ποια πρωτοβουλία θέλετε να ξεκινήσουμε για να μεταδώσουμε ευρωπαϊκές αξίες σε όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης στο εθνικό επίπεδο αλλά και στα ευρωπαϊκά προγράμματα και να μην κοιτάμε μόνο τι προσόντα και τι επίπεδο θα τελειώσει ο καθένας αλλά να δούμε και την ψυχή αυτή της Ευρώπης γιατί συχνά το ξεχνάμε. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν λίγο περισσότερη προσοχή σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Σαμπίν για αυτό, τα σημαντικά ζητήματα που τόνισες. Θα δώσω το λόγο τον κύριο Γραμματικάκη και μετά Μακλάρκιν πρώτο ο κύριο Γραμματικάκης και μετά εσείς. Παρακαλώ κύριο Γραμματικάκη νομίζω κυρία Πρόεδρε ότι είναι σημαντική η σημερινή μέρα. Η εισαγωγή σας πρώτα-πρώτα έδειξε το πλούσιο έργο της Επιτροπής Πολιτισμού και θα έλεγα ειδικά τον τελευταίο χρόνο παρά τις δυσκολίες που βρίσκεται και παρά τις επιφυλάξεις που συχνά εκφράζει η επίσημη ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες που μου συμβαίνει σπάνια τις τοποθετήσεις των τριών θεσμικών εκπροσώπων, διότι είχαν ειλικρίνεια. Νομίζω ότι από το στάδιο των μεγάλων λόγων όταν περάσουμε στην ειλικρίνεια στο πόσο δύσκολο είναι τα προβλήματα, στο πόσο η γραφειοκρατία τα εμποδίζει, στο πόσο η ίδια η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα καθιστά δυσεπίλητα, διότι πολλοί πρέπει να συνεργαστούν είναι ένα πρώτο βήμα. Από αυτή όμως την εντύπωσή μου που σας λέω είναι θετική ότι υπήρξε ειλικρίνεια και από τους τρεις ομιλήσαντες, επισήμους θα τους έλεγα, η πραγματικότητα πάλι βοά. Εγώ θα πω δύο στοιχεία μόνο, ίσως αναφέρθηκαν, στην πατρίδα τη χώρα μου, την Ελλάδα, φαντάζομαι και οι άλλες χώρες απειλούνται από παρόμοια νούμερα, η ανεργία των νέων φτάνει το 51% παρακαλώ αυτή τη στιγμή, των πτυχιούχων, με στοιχεία επίσημα του 2015. Αυτό, συγγνώμη που θα γίνω πολύ προκλητικός, έπρεπε να κηρύξει για την Ευρώπη επίπεδο συναγερμού όπως στις Βρυξέλλες αυτές τις δυσίωνες μέρες πέντε, το ανώτερο δυνατόν. Δεν μπορεί η πετυχημένη Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρά προς το μέλλον με τέτοια, αν θέλετε, ποσοστά ανεργίας. Δεύτερο και πάρα πολύ χαρακτηριστικό σε όσα αξιόλογα είπατε. Ε, το 1 τρίτο νομίζω το ανέφερε ο κύριος Επίτροπος είναι ακριβές, 28% λένε τα δικά μου νούμερα, το 1 τρίτο περίπου των νέων ψήφισε στις τελευταίες εκλογές. Παρόλα αυτά, με επίσημες θα έλεγα υπολογισμούς, δημοσκοπήσεις, το 75% των νέων είναι υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει μια μεγάλη απόσταση από τα θεσμικά μας όργανα και θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ευθύνη. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι θέλουν την Ευρώπη, ας το πω έτσι χοντρικά, αλλά από την άλλη μεριά δεν ενδιαφέρονται για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα. Δύσκολα λοιπόν και δυσεπίλητα προβλήματα. Γίνονται πολλά, υπάρχουν καλές προθέσεις, αλλά φοβούμαι ότι δεν είναι αρκετά και τις ταλαιπωρίες που υφίσταται ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα το Έρασμος νομίζω θα μπορούσαμε να τους αποφύγουμε. Τι λείπει λοιπόν. Το υπονοήσατε μερικοί, εγώ θα το πω πιο ανοιχτά. Ένα πραγματικό όραμα για τους νέους. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Δεν αρκεί μόνο να καταπολεμηθεί η ανεργία, δεν αρκεί καθόλου ο συντονισμός, δεν αρκεί να αλλάξουν οι δομές. Σε τελευταία όμως ανάλυση και θα σας εκπίξει Είμαι αισιόδοξο. Και ο λόγο είναι πάρα πολύ απλό. Can you conclude please because yes, have... yes, okay. yes. Είπα ότι είμαι αισιόδοξο και ο λόγο είναι πολύ απλό. Οι αξίε που στηρίζεται αυτό το μεγάλο πείραμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δοκιμαστεί και είναι αιώνιε. Και αυτή τη φορά με τη συμπαράσταση που δείχνουμε όλοι στους Γάλλους αυτές οι αξίες θα υπερισχύσουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Grazie. Pregherei tutti di rispettare Ευχαριστώ. Παρακαλώ όλους τους αγορητές να τηρήσουν το χρόνο μιλίας τους. Θα δώσω τηλέφωνο, στο, λόγο συγγνώμη στην κυρία Μακλάρκιν και μετά στον κύριο Δημήτρη Μπαξεβανάκη. Uh, um, Ευχαριστώ και καλώς ορίζω όλους τους ε, καλεσμένους μας που ήρθαν από άλλα κοινοβούλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολο να έρθει κανείς Βρυξέλλες και βεβαίως προξενεί και ανησυχία. Τα σου ευχαριστώ λοιπόν που ήρθαν. Ήθελα να πω πως η Επιτροπή μας είναι η φωνή των νέων και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τους στηρίξουμε στην πορεία τους και ελπίζω να ακουστεί και η φωνή τους μέσα τους δουλειά που κάνουμε. Και χαίρομαι που τόσοι πολλοί εδώ πέρα ακριβώς ε, είναι από το Φόρουμ των Νέων. Είναι χρήσιμο ακριβώς ε, όταν μιλάμε για τα προβλήματα της ε, ριζοσφαστικοποίησης να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μέσω της εκπαίδευσης. Και εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια στο Ηνωμένο Βασίλειο πήγα σε έξι διαφορετικά σχολεία στην περιφέρειά μου σε μια ημέρα της Δημοκρατίας και οι νέοι αντιδρούσαν ε, στο να κολλάμε ετικέτες για το ότι συγκεκριμένες μέρες του πληθυσμού ε, τις ε, ξεχώριζαν και τις περιθεροποιούσαν και το θεωρούσαν ως μια επίθεση στους νέους γενικά. Ότι ήταν μια επίθεση σε όλους τους νέους. Το ενδιαφέρον είναι ότι ήθελαν να μάθουν περισσότερα, ήθελαν να καταλάβουν τις διαφορές για να ρίξουν μόνο τους τους τύπους. Αλλά οι δάσκαλοι μου είπαν ε, εμείς θα θέλαμε να μάθουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τους δασκάλους μας ε, να βοηθήσουν τους ε, νέους να δουν όλες αυτές τις μεγάλες ιδέες και θα ήθελα να φέρω κάτι για την διαβίω εκπαίδευση κτλ. Μιλάμε συνεχώς για το Εράσμος και την επιτυχία του. Θεωρώ πως τώρα πρέπει να εστιάσουμε στη διαβίω εκπαίδευση και τα επαγγελματικά προσόντα και το πώς μπορούν να βοηθήσουν τους νέους που ίσως έμειναν πίσω να τους ε, δώσουν μια διαφορετική πορεία και πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να τους στηρίξουμε, να στηρίξουμε τους ε, δασκάλους μας ε, στη μάχη κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Πώς μπορούμε τώρα να εστιάσουμε περισσότερο στους ε, θεσμούς εκείνους τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την δεύτερη ευκαιρία θα έλεγα. Σας ευχαριστώ πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον στον κύριο Δημήτρη Μπαξεβανάκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε τα δεδομένα που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του για την κατάσταση στη χώρα μου, στην Ελλάδα σήμερα, είναι οι πολιτικές λιτότητας, η ανθρωπιστική κρίση και η διάλυση της αγοράς εργασίας. Στην εξαετία 2009-2015 η μείωση της χρηματοδότησης στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανήλθε σε ποσοστό 36%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία 25.000 κενών θέσεων δασκάλων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ανεργία αποτελεί σήμερα το οξύτερο πρόβλημα στη χώρα μου. Το ποσοστό της είναι καθυλωμένο στο 26%, ενώ για τους νέους κάτω των 25 ετών, όπως ανέφερε και ο κύριος Γραμματικάκης, υπερβαίνει το 50%. Οι παρεμβάσεις στην οργάνωση της εργασίας με υποτιθέμενο στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας οδήγησαν στη διάλυση της αγοράς εργασίας. Τέτοιες παρεμβάσεις ήταν οι δραστικές μειώσεις μισθών, η επέκταση της ευέλικτης απασχόλησης, η διευκόλυνση των απολύσεων, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σε ένα τέτοιο τοπίο, κάθε προσπάθεια για προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι απλώς χωρίς νόημα. Με βάση τα παραπάνω, επιβάλλεται μια συνολική αναθεώρηση των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων με προϋπόθεση τον τερματισμό της λιτότητας που έχει επιβληθεί στη χώρα μου από τους θεσμούς μεταξύ των οποίων δυστυχώς είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επίσης δυστυχώς αγνοεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η λιτότητα πρέπει να τελειώσει. Η λιτότητα σκοτώνει την Ελλάδα, σκοτώνει την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Thank you so much. And now I give the floor to Mrs. Ο λόγος στην κυρία και μετά θα περάσουμε ξανά σε εκπροσώπηση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσουμε για την εκπαίδευση και την νεότητα με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων καθώς επίσης και με τους νέους που εκπροσωπούνται εδώ μέσω του Youth Forum. Σε αυτό το επίπεδο θα ήθελα να σας μιλήσω για τον διασωτικό διάλογο των τελευταίων 18 μηνών που βοηθάει την, στην συμμετοχή των νέων στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υποβάλουμε, να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα αυτού του διαλόγου που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πιστεύω ότι αυτά τα συμπεράσματα μπορούν να συνεισφέρουν για να ε, ε, σχεδιάσουμε καλύτερα την πολιτική για την νεότητα και να αναπτύξουμε την εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη τους νέους. Στην Επιτροπή μας ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τον διάλογο με τους νέους και ε, ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που άκουσα τις ε, παρουσιάσεις ε, αυτές των προγραμμάτων για την νεότητα. Μισό λεπτό γιατί έχουμε έναν κατάλογο προσώπων η κυρία Φρανζέσκα Πουλίζη και μετά Νέκοφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτή την ευκαιρία διαλόγου που μας παρέχεται. Η χώρα μου, η Ιταλία, αντιμετωπίζει μια σκληρή διαδικασία μεταρρυθμίσεων προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη στοχεύοντας ε, πρώτα απ' όλα στην ε, εκπαίδευση. Έχουμε ένα τραγικό ποσοστό ανεργίας των νέων που ξεπερνά το 40%. Έχουμε ένα ποσοστό εγκατάλειψης των σχολιών, ε, που σήμερα βρίσκεται στο 17% αλλά πέραν από τους στόχους της ευρωπαϊκής σύγκληση που πρέπει να πετύχουμε έχουμε και στόχους ε, εσωτερικής σύγκληση ε, που θα πρέπει να αποκαταστήσουμε για να προσφέρουμε σε όλους τους νέους και τις νέες ίσες ευκαιρίες. Αγόρια και ε, κοπέλες που ζουν στο νότο της Ιταλίας και βρίσκονται στο ποσοστό του 26% σε ό,τι αφορά την εγκατάλειψη των σχολείων, ενώ στον Βορρά έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά, αν και εκεί υπάρχουν ε, διαφορές ανάμεσα στις ε, ε, μετροπολιτικές περιοχές και τις υπόλοιπες. Για να πετύχουμε λοιπόν αυτούς τους στόχους προσπαθούμε καταρχήν να εισαγάγουμε το διαδικό σύστημα στο σύστημα εκπαίδευση, αλλά θα πρέπει να αυξήσουν σε σχέση με τις περικοπέ των παρελθόν τον αριθμό των ε, νηπιαγωγείων. Και το ερώτημά μου προς τον Επίτροπο είναι πώς να βοηθήσουμε τα κράτη που βρίσκονται σε μια θέση εάν ε, συνεχίσουν να υπολογίζονται οι δαπάνες για την εκπαίδευση στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας. Πρέπει να αφαιρέσουμε τις ε, ε, επενδύσεις αυτές από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ενδιαφέρουσα η πρόταση, όχι επειδή προέρχεται από την Ιταλία, αλλά επειδή την ε, συμμερίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Κυρία Νέκοφ, έχει το λόγο. Ο κύριος, συγγνώμη, Σας ευχαριστώ. Άκουσα όλες τις ε, παρεμβάσεις, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Εγώ θα ήθελα να φερθώ σε αυτά τα οποία είπε το Φόρουμ της Νεολαίας. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ είμαι εισηγητής ε, των σοσιαλιστών για το ίδιο θέμα. Το πρώτο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι δεν υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ της στρατηγικής των νέων και των άλλων στρατηγικών. Παραδείγματος χάρη, η στρατηγική για την εκπαίδευση του 2020 δεν αναφέρεται καθόλου το ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό γιατί η εκπαίδευση πρέπει να είναι στη, βάση της στρατηγικής μας για την νεολαία. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την ε, στήριξή μου. Στις 16 Νοεμβρίου είχαμε μία συζήτηση στρογγυλή τραπέζη για να συζητήσουμε αυτά ακριβώ τα ζητήματα και χτε μιλήσαμε και για την διαβίου κατάρτιση. Όλα αυτά τα φόρουμ πρέπει να επικοινωνούν. Και καλωσορίζω την πρωτοβουλία να δημιουργηθεί μια άτιμη πλατφόρμα διαβίου κατάρτισης. Μιλήσατε για το 50% οι οργανώσεις ε, της νεολαίας κατά 50% θεωρούν πως ε, δεν λαμβάνονται υπόψη αυτά τα οποία λένε στην πολιτική για τους νέους. Θεωρώ πως η φωνή των οργανώσεων της νεολαίας ε, πρέπει να ακουστεί. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και σας διαβεβαιώ πως όλες αυτές οι συστάσεις θα εμφανιστούν στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστώ και παρακαλώ λοιπόν και τους ε, σκιώδεις εισηγητές να έρθουν σε επαφή μαζί σας για να υπάρχει ακριβώς μια συνέχεια στον δομημένο διάλογο με το Φόρουμ της Νεολαίας. Τώρα λοιπόν... Δώσω το λόγο στην κυρία Γιάνγκ από την Αυστρία. Ε, Η Αυστρία έχει μεγάλη παράδοση στο διπλό σύστημα εκπαίδευσης ε, επαγγελματικής ε, και μη. Το ζήτημα λοιπόν ε, είναι τι κάνουν οι χώρες που δεν έχουν μια τέτοια παράδοση για να επεκτείνουν ακριβώς το εκπαιδευτικό του σύστημα. Εμείς με το σύστημα αυτό έχουμε πολύ χαμηλή ανεργία των νέων η οποία βεβαίως εντάξει λόγω της οικονομικής κρίσης είναι 12% είναι πολύ υψηλή παρόλα αυτά για το τι έχουμε συνηθίσει. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω και το εξής. Ε, είδα και πρόσεξα από ε, τις διαφορετικές πληροφορίες που δώσατε και σας ευχαριστώ για αυτό. Δεν ακούστηκαν κάποια πράγματα. Το ένα είναι η οικογένεια, οι αξίες και οι επιδόσεις. Ε, και το ερώτημά μου είναι Πώς εντάσσονται αυτά στην στρατηγική σας. Ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, δεν εφήγησαν όλα τα ζητήματα στις παρουσιάσεις, αλλά νομίζω πως αυτά που ακούσαμε είναι ιδιαίτερα σημαντικά και θεμελιώδη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τον Λουίτζι Μόργανο, τελευταίος παρεμβαίνων και μετά θα δώσουμε το λόγο στους ε, είναι γνωστές οι αρμοδιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα παιδείας, ε, εκπαίδευση κλπ. Λοιπόν, η σημαντική συνάντηση από εκεί ξεκινάει και προτίθεται να προσεγγίσει τις συνολικές στρατηγικές, κάτι το οποίο συχνά όλοι τονίζουμε. Αλλά είναι προφανές πως και εδώ η πολιτική θα πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο της. Γίνεται αναφορά στην Κομισιόν, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή, αν αυτά τα οποία γίνονται για τα σχολεία, το πανεπιστήμιο, την πανεπιστήμια κατάρτιση αποτελούν επένδυση, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το θεωρούμε ως δαπάνη. Το πολιτικό αίτημα είναι ακριβώς αυτό, διότι σε αυτούς τους κλάδους απαιτούνται πόροι, όπως είπε ήδη η γερουσιαστής που το ζήτημα του Συμφώνου Σταθερότητα επί του θέματος αυτού δεν μπορεί να τεθεί στο ίδιο επίπεδο με άλλε ε, επαρεμβάσεις. Γνωρίζω ότι όλοι μπορούν να πούνε ότι ο καθένα έχει τι ανάγκε του, αλλά αν δεν είμαστε κανένα να δώσουμε προτεραιότητα, τότε η ευθύνη καθενό μα ε, εξαρτάται από τις πράξεις του. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα και εγώ να τονίσω αυτή την επιτυχία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από καιρό έχει θίξει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του ταμείο, ταμείου δηλαδή να αποκλειστούν όπως αποκλείονται από τα διορθωτικά ταμεία και από τη συγχρηματοδότηση οι δαπάνες για επενδύσεις, να θεωρηθεί η εκπαίδευση ως επένδυση και να αποχωριστεί από τον, ε, τον κανόνα αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρομαι στο ρόλο που είδαμε στο Κοινοβούλιο για το ζήτημα Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, Υπουργό, στον Επίτροπο και στο Youth Forum για τις ε, απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κάποια λόγια για τις ε, διάφορες παρεμβάσεις που ακούσαμε. Επανειλημμένα συστήθηκε ότι δεν χρειάζεται να στοχεύουμε την εκπαίδευση, δηλαδή το, τυπικό σύστημα εκπαίδευσης ε, για την καλύτερη ένταξη των μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία αλλά και το άτυπο την μορφή εκπαίδευση. για αυτό το λόγο και η Λουξεμβουργική Προεδρία πρότεινε οι τη διατάξει περίπου ταυτόσιμε για την ε, συνεδρίαση του Συμβουλίου Νεότητας ε, και του Συμβουλίου Εκπαίδευση και είτε πρόκειται για νέους πρόσφυγες ή μετανάστες που ήρθαν τώρα με την κρίση ή που είχαν φτάσει στην επικράτειά μας εδώ και μερικά χρόνια και να προκύψουν τα προβλήματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο στο Συμβούλιο Εκπαίδευση που συζητήθηκε το ζήτημα, αλλά και στο Συμβούλιο Νεότητας ε, Νομίζω πως η πολιτική συμμετοχή των νέων ε, είναι θέμα πολύ σημαντικό, διότι φυσικά η επιτυχία στο σχολείο το να αποκτήσει ένα, ένα απολυτήριο και στη συνέχεια ε, είναι πολύ σημαντικό για την ένταξη στην κοινωνία και στην ενεργοζωή. Αλλά θα πρέπει να είσαι και πολίτης ε, με πλήρη δικαιώματα ένας πολίτης ο οποίος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει και να εκφράσει τη γνώμη του και ενδεχόμενα να αλλάξει κάποια πράγματα που δεν του αρέσουν στις κοινωνίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε την περιθωριοποίηση πολλών νέων και φυσικά να αποφύγουμε τον κίνδυνο της ριζοσπαστικοποίησης. Αυτά ιδιαίτερα ήθελα να τονίσω. Θεωρώ ότι πολλές από τις προτάσεις που ακούστηκαν καταρχήν δεν είναι καινούργιες, Συζήτησαμε για το Erasmus Plus, συζήτησαμε για την επέκταση του Erasmus Plus, πώς μπορούμε να ε, το διευρύνουμε σε άλλους τομείς από τους παραδοσιακούς όπως ανταλλαγή φοιτητών ε, ανάμεσα σε διάφορες χώρες. που έχει ιδιαίτερη σημασία για να εκδημοκρατιστεί το σύστημα του Erasmus Plus. Αλλά και επανερχόμεθα στο ζήτημα των βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη, όταν πρόκειται για το ε, θέμα της διτής εκπαίδευσης, ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να ενταχθούν καλύτερα οι μεταναστες οι ή πρόσφυγες. Υπάρχουν κράτη-μέλη στην, Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργούν αποτελεσματικά σε αυτά τα ζητήματα της ένταξης. Που... Και εδώ ε, και αυτό μπορεί ε, να, επιτευχθεί με την ανταλλαγή των πρακτικών. Δεύτερον, πολλά υπόθηκαν σχετικά με το σύμφωνο σταθερότητα και τα μέσα τα οποία υπάρχουν για να επενδύσουμε περισσότερο σε μια ε, ενεργό συμμετοχή των νέων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Γνωρίζουμε τους περιορισμούς που επιβάλλονται πρώτα απ' όλα από τις δημοσιονομικέ ανάγκες αλλά και από του ευρωπαϊκού μηχανισμού. Δεν νομίζω ότι σήμερα σε αυτή τη συνάντηση ή σε ένα Συμβούλιο Υπουργών εκπαίδευσης ή νεότητας ε, να αλλάξει το όλο σύστημα. Ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω για μια ακόμα φορά την πρόταση της Λουξεμβουργικής Προεδρίας για μια παρέκκληση όλων των δαπανών που τώρα είναι απαραίτητε ε, για την ένταξη των προσφύγων και για τη συμμετοχή τους στα συστήματά μας και να μην καταχωρούνται στα συστήματα όπως γίνονται τώρα. Έτσι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε ή να ε, μην κάνουμε κάποιες επενδύσεις από άλλους ε, κλάδους του προπολογισμού. Αυτό δεν πρέπει να γίνει διότι θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δώσουμε τώρα τα μέσα σε όλα τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να αντιδράσουν και να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που είναι πολύ σοβαρή αλλά και πολύ επικίνδυνη για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Δίνω το λόγο τώρα στον Επίτροπο, κύριο Ναυράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να χωρίσω δύο τμήματα την απάντησή μου τη διάγνωση και τη θεραπεία, διότι συμφωνώ με τους εκπροσώπους των ε, κοινοβουλίων που υπογράμμισαν τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. Ε, ορισμένες δημοσιονομικές ε, πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη-μέλη συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι η νεολαία και η εκπαίδευση μπορούν να είναι, είναι πιθανό να αποτελέσουν το πιο σημαντικό θύμα των δημοσιονομικών αυτών πολιτικών. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, είναι και κατά κάποιο τρόπο κατανοητό ότι οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να ε, ίσως καλέσουν τους ε, προϋπολογισμούς τους και να κάνουν περικοπές για να γίνει πιο, για να εξηγιανθεί η οικονομία. Όμως ε, οι πολιτικές αυτές, οι δημοσιονομικές αυτές πολιτικές ε, απομείωσαν τις ε, πολιτικές που κοιτούν προς το μέλλον. Όπως είπε ο κ. Μοργάνο, οι, πολιτικέ πολιτικές για την νεολαία και την εκπαίδευση είναι ε, επένδυση στο μέλλον. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι πρέπει να επενδύσεις σήμερα και να δεις τα αποτελέσματα αργότερα. Είναι πολύ δύσκολο να πείσει ε, αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις και σχεδιάζουν τις πολιτικές σήμερα να επενδύσουν στο μέλλον διότι το μέλλον πολύ συχνά ξεπερνά τις εκλογικές προθεσμίες ε, και οι πολιτικοί θέλουν αυτά αποτελέσματα πριν τις επόμενες εκλογές. Θα πρέπει όμως να τους πείσουμε ότι η εκπαίδευση είναι αξιόλογη επένδυση και όχι μόνο αυτή καθεαυτή ο, αλλά και ως επένδυση για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, για την ε, αύξηση της συνοχής της κοινωνίας και για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση. Και έχουμε μέσα για να ε, χαρτογραφήσουμε την κατάσταση σήμερα. Έχουμε την έκθεση για την νεολαία, έχουμε ε, το στρατηγικό πλαίσιο πέρσι κατάσταση 2020, έχουμε τις αιτήσεις εκθέσεις αξιολόγησης, Οπότε βλέπουμε τάση βελτίωσης και έχουμε ελπίδες να πετύχουμε τον βασικό μας ε, στόχο για την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου μέχρι το 2020. Επίσης για τον στόχο ε, της ε, ε, λήψης πτυχίου από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέχρι το 2020. Όμως αντιμετωπίζουμε και σοβαρές δυσκολίες και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσα μέσα διαθέτουμε, όχι μόνο το έρασμος συν αλλά και την εγγύηση για την νεότητα, την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ε, αλλά και ε, εργαλεία της πολιτικής απασχόλησης και της πολιτικής εκπαίδευσης ταυτόχρονα και παράλληλα. Για να γυρίσω όμως τώρα στη θεραπεία. Το Erasmus Plus είναι προφανώς ένα πολύ βασικό πρόγραμμα ε, του χαρτοφυλακίου μου και αφορά την κινητικότητα των ε, ε, φοιτητών αλλά έχουμε και πρόγραμμα κινητικότητας των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνικών γυμνασίων και ηλικίων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα κινητικότητας του Erasmus Plus, ε, να τους δώσουμε την ευκαιρία να επισκεφτούν μια άλλη χώρα, να αποκτήσουν γνώσεις για μια άλλη εταιρεία, μέσω μαθητείας κλπ. Είναι μια καλή αρχή για αυτούς που βρίσκονται ε, σε, στα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε όμως και τα προγράμματα e-training, ηλεκτρονικής κατάρτισης, που φέρουν σε επαφή σχολεία και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ε, σχολεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν συμμετοχές, ε, και από σχολεία που δεν αποτελούν από σχολεία που δεν βρίσκονται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ευρώπη και από την Αφρική. Οπότε αυτή η ηλεκτρονική κατάρτιση δημιουργεί σχέση μεταξύ σχολείων και μαθητών ε, και φοιτητών ε, έτσι ώστε να κατανοήσουμε, να κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τον άλλον και να επικρατήσει ανεκτικότητα. Συμφωνώ για την σημασία της άτυπης ε, κατάρτισης ό,τι αφορά τη διαβίωματιση, της άτυπης εκπαίδευσης. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά μας συστήματα είναι υπερβολικά παγιωμένα και παραδοσιακά ε, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ε, του σήμερα. η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη για τους περισσότερους από αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται όλοι αυτοί να αποκτούν νέες γνώσεις ε, και νέες δεξιότητες. Είναι βασική απέτηση των καιρών. Ακριβώς εξαιτία της ε, συνεχούς αναδιάρθρωσης της οικονομίας, εξαιτία της ε, ψηφιακής επανάστασης, εξαιτία ε, της επανάστασης που λαμβάνει χώρα στον τριτογενή τρομέα κλπ. Οπότε θα πρέπει σε όλα μας τα project, σε όλα μας τα, τα σχέδια να την υποστηρίζουμε ε, να υποστηρίζουμε προγράμματα διαβίου μάθησης και άτυπη εκπαίδευση. Το ειδικό μου χαρτοφυλάκιο είναι πλατή σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του, ε, αλλά τα διάφορα συστατικά του στοιχεία μπορούν να αλληλοβοηθηθούν. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τους, ε, το μεταναστευτικό, η άθληση, το αθλητισμός μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο την ενσωμάτωση των νέων μεταναστών ή προσφύγων. Γιατί ίσως ο αθλητισμός είναι η πιο δημοφιλής ε, γλώσσα και είναι σημαντικό και πολύ καλό εργαλείο για την ένταξη όλων των κοινοτήτων προσφύγων και μεταναστών. Ε, ε, μ' αρέσει η ιδέα για το σύμβολο σταθερότητας για την εκπαίδευση, ε, αλλά υφίσταται και η αρχή της επικουρικότητας και δεν μπορώ να υιοθετήσω ένα τέτοιο ε, σύμφωνο σταθερότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόεδρος, χρειαζόμαστε καλύτερη συμμαχία μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και Κομισιόν για να πείσουμε το Συμβούλιο. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ο κ. Παλ. Γιατί έχουμε καθυστερήσει. Και μετά θα καλέσω τους επόμενους ομιλητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις με πολλές από τις οποίες ε, συμφωνώ. Κοιτάξτε, συχνά στις επιτροπές αυτές ε, έχουμε το πρόβλημα ότι τα λέμε μεταξύ μας εμείς που συμφωνούμε. Και η μεγαλύτερη πρόκληση, όπως είπε και η Ευρωβουλευτή Συνέκο, το θέμα είναι οι πολιτικές αυτές να πάνε στα άλλα φόρα και οι επιτροπές του Κοινοβουλίου και να πείσουμε και τους άλλους πως ε, όντως η εκπαίδευση είναι επένδυση στο μέλλον. Ε, νομίζω λοιπόν πως ε, το ότι είμαστε εδώ πέρα σήμερα έχουμε, είναι μια απόδειξη του ακόμα και όταν μειώνονται οι προπολογισμοί μπορούμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις ε, στους ε, νέους. Δεύτερον, η ένταξη δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο έρχεται δεύτερο. Πρέπει να είναι πιο ανοιχτά τα συστήματα της εκπαίδευσης. Ε, δεν μπορεί να λυθεί τώρα με το να γίνουν ειδικά σχολεία Πρέπει όλα μας τα σχολεία να είναι καλά στην ένταξη. Και τέλος, κάτι το οποίο ίσως λείπει από την ευρωπαϊκή πολιτική, είναι μια πραγματικά ευρωπαϊκή αντίληψη όσον αφορά την ιδιότητα του πολίτη, που θα είναι κάπως συμμετοχική. Και ακριβώς έτσι θα πρέπει να δούμε το πώς θα διδάξουμε την Ευρώπη στους νέους σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως βλέπετε οι νέοι έχουν ιδέες ε, που είναι χρήσιμες, εμπλουτίζουν το διάλογό μας, τη σκέψη μας και ε, αγαπητέ αλλά σήμερα είναι μία από τις φάσεις του διαλόγου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις εκθέσεις σχετικά με τους νέους. Είμαι βέβαιη πως ε, γίνονται συναντήσεις Βέβαια και η συνάδελφος Νέκοφ νωρίτερα, έχουμε και τον σκιώδη διηγητή σας και δεν είναι ανταγωνιστική η σχέση μας. Ολοκληρώνονται οι εργασίες μας, συμπληρώνονται και πρέπει να κάνουμε νέες πολιτικές για τους νέους και όχι πεπαλαιωμένε πολιτικές να πω ότι αυτό το οποίο συζητήσαμε και ευχαριστώ για την ειλικρίνεια των προτάσεων που έφτασαν και από τον Επίτροπο και από τον Υπουργό ότι υπάρχουν όμως σε όλα ένα όρια να το, το ξέρουμε αυτό αλλά δεν θέλω να το βάλουμε μια τελεία σε αυτό το πάνελ που είναι κάπως πιο πολιτικής φύσης δεν θα ήθελα λοιπόν όπως ανακαλύψαμε τη σημασία της ε, κληρονομικής της πολιτικής, πολιτικής κληρονομιάς να ανακαλύψουμε την ε, πολιτική ε, για την νεότητα και την εκπαίδευση μετά από τη ριζοσπαστικοποίηση και όπως ε, αυτά τα παιδιά όπως είπαν και οι δάσκαλοι στο Σαντονί είναι και δικά μας. Θα πρέπει να είναι ένας άλλος τρόπος για να δούμε τα πράγματα αλλά και η εκπαιδευτική προσέγγιση αλλά και η διαπολιτισμική προσέγγιση. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε τους κανόνες ομού με έναν πρωταγωνισμό των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που θέλουν να έχουν οι νέοι και θέλουν να μας προτείνουν. Πρέπει να αποκτήσουμε ένα εγκάρσιο μέσο για τις πολιτικές με το οποίο συζητάει το φόρουμ και είναι το ε, διακοινοβουλευτικό φόρουμ με το οποίο συμμετέχουν οι συνάδελφοι από όλες τις επιτροπές και στο οποίο συμμετείχα και εγώ στο παρελθόν όχι ως νέα ως επειδή με ενδιαφέρει το ζήτημα, νομίζω λοιπόν ότι είναι μια πολύ σημαντική φωνή με την οποία θα πρέπει να διαδράσουμε. Θα δώσω το λόγο Ε, μάλλον να ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα δύο πάνελ, να δώσω το λόγο στον Ντέιβιντ Λόπε και στον Ρομπέρτο Ρουφίνο να έρθουν εδώ στο Προεδρείο. Ο Λόπε είναι πρόεδρο για θέματα ε, διαβίου μάθηση ε, που θα μιλήσει για ένα ζήτημα το οποίο πρόκειψε από τι παρεμβάσει σα. Life Learning και ο ρόλο του Life Plus και ο δεύτερο είναι ο Ρομπέρτο Ρουφίνο ε, επίτιμος πρόεδρος ε, και γενικό γραμματέας της ε, Φοντασιόν Ιντερκουλτούρα, δηλαδή του Δήματος Ιντερκουλτούρα. για την ενεργό ηθαγένεια στο πλαίσιο του τριμηνιαίου προγράμματος. Ευχαριστώ. Allora, we start. Eh? As soon as possible, okay? Allora, we start with, uh, with uh, David Lopez, please. je vais... Καλή σας μέρα, θα μιλήσω στα γαλλικά. Το έγγραφο της παρέμβασής μου θα το βρείτε στα αγγλικά μεταξύ των εγγράφων τα οποία σας διανεμήθηκαν. Να διευκρινίσω ότι η οργάνωση είναι πλατφόρμα διαβίου μάθησης. Platform, όχι program όπως λέγεται στο έγγραφο της ημερησίας διάταξης. Έχουμε αλλάξει το όνομα εδώ και 10 χρόνια, από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε καταφέρει να ε, συνηθίσουμε στο καινούργιο όνομα. Πολλά ελέγχθησαν, ε, περί της ουσίας ε, δεν θα επανέλθω, στηρίζω πλήρω την ανάλυση του Αλαν Παλ, άλλωστε συνεργαζόμαστε με το Youth Forum και πολλές άλλες άλλωστε οργανώσεις νέων συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας. Να πω όμως ότι, να τονίσω μάλιστα ότι η εκπαίδευση δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση όπως υπόθηκε πολύ σωστά. Θα αναφερθώ στην διαβίου μάθηση, στα προγράμματα και τις τεχνικές, ε, να σας πω ότι μετά την ενδιαμεσή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εν ώψη της έκθεσης του Δεκεμβρίου 2017 και μετά την δημόσια διαβούλευση του 2014, την οποία κάναμε εμείς, ε, το καλοκαίρι του 2015 ετοιμάσαμε μια αιτήσια έκθεση για να αξιολογήσουμε τη γνώμη των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά το δεύτερο γύρο των αιτήσεων του Erasmus Plus. Συλλέξαμε 275 απαντήσεις σε τέσσερις γλώσσες. Ο στόχος της ε, ε, μελέτης αυτής ήταν να επιβεβαιώσουμε το κατά πόσον το Erasmus Plus στηρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες τις οποίες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κατά πόσον το πρόγραμμα αυτό έχει πραγματικές ε, συνέπειες σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές κοινωνίες για την ε, αλληλοκατανόηση, την κοινωνική ένταξη και την βελτίωση της, της, ε, των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της κινητικότητας. Η έκθεσή μου ε, επιβεβαιώνεται όσα είπε η στην αρχή σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή που είναι απαραίτητη να εξασφαλιστεί μέσω αυτών των προγραμμάτων. Ε, οι ερωτώμενοι εξέφρασαν πολύ θετική άποψη για το Erasmus Plus. Είναι μοναδική ευκαιρία χρηματοδότησης ε, και μάλιστα ήταν και πολλά πειράματα από το πρώτο πρόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια. Το 86% των ερωτωμένων ε, θεωρούν ότι το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ ή σχετικά ε, ε, εστιασμένο και έχει βρίσκεται σε συνάδει με τις ανάγκες και την πραγματικότητα. παρόλο ότι τα μέλη, τα, τα, μέλη μας χαίρονται για την απλοποίηση του προγράμματος μπορούν να γίνουν ακόμα πολλά βήματα. Και πρώτον, η διάσταση του, η διάσταση, ε, η, συνιστόσα δηλαδή διαβίου μάθησης του Erasmus Plus. Ε, το βασικό πλεονέκτημα του Erasmus ε, Plus είναι ακριβώς η διατομεακή του προσέγγιση και η εστίαση στην διαβίου μάθηση. Ε, συνδυάζοντας πολλά παλιότερα προγράμματα διαβίου μάθησης, Εράσμους, Λεωνάρντο Νταβίντσι, Κομένιους, Γκρούντβιχ κλπ, ε, το Youth in Action, ε, το Erasmus Mundus κλπ, μέσα κάτω από την ίδια ομπρέλα. Ο στόχος ήταν ακριβώς να υπογραμμιστεί αυτή η διάσταση διαβίου μάθησης. Και ο χωρισμός του προγράμματος σε κλειδιά θα έπρεπε να αποτελέσει εγγύηση για αυτήν την καινούργια προσέγγιση. Στην πράξη, πιστεύουμε ότι ε, είναι δύσκολο να υλοποιηθεί αυτή η ομπρέλα δεδομένου ότι ο καθένας παραμένει στον τομέα του. Πολύ συχνά οι εθνικές υπηρεσίες ή και η Ευρωπαϊκή ε, Αρχή ε, δεν αξιολογεί ορθά τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν το καθένα από το πλαίσιο τους. Για παράδειγμα, μας δόθηκε ένα από τα μέλη μας. Αν θέλετε να υποβάλλετε ε, ένα έργο για την κατάρτιση των γονέων. Ε, ένα τέτοιο, ένα τέτοιο πρόγραμμα εστιάζει και στην άτυπη εκπαίδευση των γονέων αλλά και την εκπαίδευση των παιδιών και των νέων. Δηλαδή έχει διπλό κοινό. Δυστυχώς όμως αυτό το πρόγραμμα πιθανώς θα απορριφθεί γιατί, γιατί σε ορισμένες χώρες οι αξιολογητές, ορισμένοι αξιολογητές θα θεωρήσουν ενδεχομένως ότι αφεν, ε, ότι απευθύνεται πιο πολύ στους γονείς ενώ κάποιοι άλλοι ότι απευθύνεται πιο πολύ στα παιδιά με αποτέλεσμα να δώσουν αρνητική αξιολόγηση θεωρώντας ότι το έργο, η πρόταση αυτή είναι υπερβολικά πλατιά ή υπερβολικά σαφής. Αντιθέτως, άλλοι αξιολογητές μπορεί να θεωρήσουν ότι το πρόγραμμα αυτό αξίζει σηματοδότησης. Νομίζω λοιπόν ότι ε, υπάρχουν εμπόδια στην ανάπτυξη διατομεακών σχεδίων και έργων. Ενθαρρύνουμε λοιπόν την Κομισιόν να ε, ε, υποστηρίξει τέτοια προγράμματα και να επιμείνει στην υποστήριξή τους ε, και κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων κατάρτισης των εθνικών αξιολογητών και κατά τη διάρκεια των ημερίδων εφαρμογής και υλοποίησης. Δεύτερο, δεύτερο σημείο. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις δράσεις τις, μάλλον σε ό,τι αφορά την ε, δράση κλειδί υπαριθμών 3. Έχουμε 39 δίκτυα ως μέλη και το καθήκον τους, η αποστολή τους είναι διπλή. Αφενός ε, να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές προς τα κάτω, σε τοπικό δηλαδή επίπεδο, με ανταλλαγή καλών πρακτικών, αλλά και από κάτω προς τα πάνω για να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, σχεδιάσει καινούργια προγράμματα για το μέλλον. Ορισμένε φορέ έχουμε την εντύπωση ότι δεν μας χρησιμοποιούν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπογραμμίζουμε ότι υπάρχει έλλειψη σε ό,τι αφορά την μεταφορά καινοτομία. Ε, το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή κάνει προσκλήση ε, ε, κάθε δύο χρόνια και πολύ περιορισμένο προπολογισμό. Έχουμε 4 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίους οι οποίοι εποφελούνται από την κινητικότητα, αλλά το θέμα είναι και η ποιότητα. Θα πρέπει να εργαστούμε και, σε, και στο θέμα της ποιότητας. Τρίτον, ναι, τελειώνεται αν θέλετε λέει η πρόεδρος, ε, οργανώσεις που βασίζονται στις Βρυξέλλες. Τι πρέπει να κάνουν, όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να γίνει αποκέντρωση του προγράμματος, Δηλαδή, ο καθένας θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει τις αιτήσει στη γλώσσα του, αλλά οι <laughs> οργανώσεις που βρίσκονται στο Βέλγιο ε, πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε γλώσσα του Βελγίου. Αυτό είναι πρόβλημα, εντάξει, λύνεται τελευταία, αλλά είναι ένα δευτερόμενο πρόβλημα, αλλά πρόβλημα. Ε, συμπέρασμα, ε, το Erasmus Plus είναι εξαιρετικό πρόγραμμα, πολύ καλό εργαλείο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διάσταση διαβίου σε αυτό διότι θα έχει πολλαπλησιαστικό αποτέλεσμα και για την κοινωνική διάσταση και για την απασχόληση και για την ε, διαπολιτισμική κατανόηση. Θα πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο της ε, δήλωσης του, των παρεσίων και είμαστε ε, διατεθειμένοι και πρόθυμοι να εργαστούμε και με την Κομισιόν και με τη Δική Επιτροπή με οποιοδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε την χαρά να βρίσκεται ανάμεσά μας κύριε Αγκαλιάτσο υπεύθυνη για το Erasmus Plus και μετά αν θέλετε να λάβετε το λόγο ευχαρίστως. Θα είναι τα λόγια μας. Θα δώσω το λόγο στον Ρομπέρτο Ρουφίνο και παρακαλώ λίγο πιο σύντομος από τον προλαλήσαντα. Κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί φίλοι, κυρίε και κύριοι. Από λίγο λόγια για ένα πρόγραμμα που λέγεται το Ευρωπαϊκό Τρίμηνο για τους πολίτες, το οποίο προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Διαπολιτισμική Μάθησης σε ένα δίκτυο θελοντών σε 24 χώρες στην Ευρώπη και ανήκει στο διεθνές πρόγραμμα AFS που ίσως έχετε ακούσει υπάρχει σε όλο τον κόσμο, ξεκίνησε πριν από 100 χρόνια, είχε ξεκινήσει με ασθενοφόρα στο, στον πόλεμο και τώρα προωθεί ανταλλαγές μεταξύ σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό για την ιδιότητα του πολίτη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το 2006 μετά από ένα πιλωτικό έργο που κάναμε εδώ με την Κομισιόν. Σήμερα περιλαμβάνει 250 Ευρωπαίους μαθητές από 20 τόσες χώρες. Κρατάει τρεις μήνες, οι μαθητές πάνε και ζουν και πάνε σχολείο σε άλλη χώρα με μια άλλη οικογένεια και έτσι ζουν πλήρως στον πολιτισμό της άλλης χώρας και στο τέλος του προγράμματος που ήταν αυτή τη βδομάδα μάλιστα συμμετέχουν σε μια πανευρωπαϊκή συνάντηση που γίνεται στις Βρυξέλλες και συζητάνε τις εμπειρίες τους πριν επιστρέψουν στις χώρες τους Λοιπόν, αυτό το κοινό σημείο των διαφόρων σημείων του προγράμματος είναι μια φάση προετοιμασίας όπου εξερευνούν μαθητές εαυτούς, τον πολιτισμό τους, την ταυτότητά τους πριν πάνε στο εξωτερικό. Υπάρχει μια φάση όπου μαθαίνουν πρώτα απ' όλα πώς ε, μαθαίνουν ε, ασχολούνται με την ξένη γλώσσα. Χτες μιλούσα με μια Ρωσίδα που πήγε στην Πορτογαλία, παραδείγματος χάρη, και δεν μιλούσε Πορτογαλικά πριν πάει αλλά είναι φοβερό το ότι μαθαίνει κανεί ε, σε τρει μήνε σε αυτή την ηλικία. Είχε μάθει και μιλούσε πορτογαλικά. Κάνουν φίλου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η συναισθηματική πτυχή δηλαδή. Έχουν μια οικογένεια που τους φιλοξενεί με αγάπη και στου τρει μήνε από το περιθώριο περνάνε να είναι μέρος της κοινότητας σε αυτή την χώρα και βλέπουν βέβαια τις διαφορές και τις ομοιότητες ανάμεσα στη δική τους χώρα και την άλλη χώρα και μετά επιστρέφουν στη χώρα τους και τα μοιράζονται αυτά με τους συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους. Εάν δούμε λοιπόν τις βασικές δεξιότητες για διαβίου κατάρτιση που έχει αναπτύξει εδώ το Κοινοβούλιο, βλέπουμε πως τουλάχιστον πέντε από αυτές έχουν άμεση σχέση με το πρόγραμμά μας. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, να γνωρίζει κανείς πώς να μαθαίνει, κοινωνικές και πολιτικές ε, δεξιότητες, ε, πρωτοβουλία και πολιτισμική έκφραση. Και βεβαίως υπήρχε μια χάρτα του Κοινοβουλίου για την κινητικότητα των μαθητών και βλέπουμε πως αυτά τα οποία αναφέρονται στη χάρτα αυτή είναι όλα σημαντικό τμήμα του τριμήνου αυτού. Ένα ε, στα άλλα σημεία που βλέπετε θα ήθελα να τονίσω δύο που έχουν για μένα μεγάλη σημασία. Το ένα είναι το ότι πηγαίνει κάποιος και έχει συμβούλους και αναγνώριση. Δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει κάποια στήριξη σε όλη αυτή την εμπειρία, να σε βοηθήσει κάποιος να αναλύσει τον πολιτισμό σου και τον άλλον πολιτισμό και βεβαίως να υπάρχει και αναγνώριση από το σχολείο, γιατί η Κομισιόν έχουμε πρόβλημα με τα σχολεία της Ευρώπης, το θεωρούν χάσιμο χρόνο. Αυτό μου λέγαν όλοι χτες, ε, γιατί λέγαν όλοι ότι θα πάω τη Δευτέρα σχολείο και οι δάσκαλοι θα μου πούνε τι, τι έμαθες στη Φιλανδία σε τρεις μήνες, τι μπορείς να μάθεις. Και το δεύτερο στοιχείο είναι το ότι ε, έχουμε όπως σας είπα αυτή την τελική συνάντηση στις Βρυξέλλες που μοιράζονται τις εμπειρίες τους ε, και σκέφτεται τι μπορούν να εφαρμόσουν στη δική τους κατάσταση και μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. δεν έχω χρόνο να τα αναπτύξω όλα αυτά. Είναι αποτέλεσμα έρευνας που κάναμε πριν από 25 χρόνια και βλέπουμε τα διάφορα επίπεδα μάθησης ε, που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της παραμονής ε, στο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη έρευνα του Μιτσχάμερ είχε γίνει από λίγα χρόνια και αν τα συγκρίνετε όλα αυτά με την μελέτη για τους ενεργούς πολίτες που είχε βγάλει η Γενική Διεθνής Εκπαίδευσης τονίζουν το ότι η αγωγή του πολίτη δεν είναι μόνο δημοκρατία, αστικά δικαιώματα κτλ. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας, με το σεβασμό, με την αντίληψη του δικού σου πολιτισμού, με το να μάθει κανείς για τον πολιτισμό και να μάθουμε πρώτα απ' όλα, θεωρώ εγώ, με το μυαλό και με την καρδιά. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν πάει κανείς σε άλλη χώρα. Δεν μαθαίνει μόνο με το μυαλό, αλλά με την καρδιά. Γι' αυτό έχει ακριβώς μεγάλη αλλαγή αυτό και μόνιμη αλλαγή στα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ μαζί σας πως ε, καμιά φορά οι δάσκαλοι λένε πως ε, αυτά είναι χάσιμο χρόνο αλλά αυτό ακριβώς ε, συζητάμε να υπάρχει μεγαλύτερη ενσωμάτωση στα διδακτικά προγράμματα Τη επίσημη και άτυπη εκπαίδευση. Λοιπόν, όπω σα υποσχέθηκα θα δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαία, αλλά πέντε ε, συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Έχουμε μόνο 30 λεπτά στη διάθεσή Θα πρέπει να παραμείνετε εντός του χρόνου που σας έχει δοθεί. Χρησιμοποίησαμε Μάλλον συγγνώμη, έχουμε 12 λεπτά, όχι 30. 12 λεπτά. Η Λουσίλη Ρία έχει το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Από το μπρος για καθέναν που θα το λόγο, το Youth Forum. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσω, να σας πω ότι έχουμε πολλούς ε, νέους εδώ και ελπίζω ότι θα βρείτε χρόνο να τους μιλήσετε και αυτοί θέλουν πολύ να σας μιλήσουν. Ε, σε ό,τι αφορά την πολιτική νεολαία, υπάρχει ένα εργαλείο, το οποίο αναφερθήκαμε άλλωστε, προκειμένου οι νέοι να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, που είναι ο διαρθρωμένος διάλογος. Και ε, θα ήθελα όλα τα μέλη των εθνικών και ιδίω κοινοβουλίων να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο, να το καταναλάβουν και να επιτρέψουν στους νέους να συμμετέχουν στο σχεδιασμό των εθνικών πολιτικών. Στον τελευταίο κύκλο που μόλις τελείωσε στο Λουξεμβουργό προέκυψε μια ιδιαίτερη σύσταση σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση του πολίτη στα, ως μάθημα στα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Θα πρέπει μάλιστα να συνεργαστούν μεταξύ τους οι οργανώσεις των νέων μαζί με τις ε, αρχές που των, της ε, επίσημης εκπαίδευσης που ρυθμίζουν τα της επίσημης εκπαίδευσης έτσι ώστε να διενεργηθούν δραστηριότητες αγωγής του πολίτη. Νομίζω ότι ανταλλάσσοντας παιδαγωγικά εργαλεία και μέσω της ε, κατάρτισης των εκπαιδευτών για θέματα αγωγής του πολίτη μπορούμε να, πετύχουμε πολλά πράγματα. Σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus Plus, ελπίζουμε ότι θα συμμετάσχει και το Youth Forum μαζί με την Επιτροπή Καλτ, γιατί έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το θέμα. Δίχως άλλο, θα αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία ως Επιτροπή για την έκθεση αυτή, αλλά θα φροντίσουμε να συμμετέχουν και νέοι. Τώρα, επτά είναι εγγεγραμμένοι. Ένα λεπτό έκαστος παρακαλώ. Θα χρησιμοποιήσω το σφυράκι μου που συνήθως το αποφεύγω. Αλλά θα το χρησιμοποιήσω κατά ημών με ύψιλον. Ο Μίκελ Ράουτ από την Εστονική Βουλή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Erasmus Plus παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Τομείο γιατί επιτρέπει στους, το γιατί επιτρέπει στους νέους ε, να κάνουν ανταλλαγέ σε ένα άτυπο περιβάλλον ε, και επιτρέπει στους νέους να εφαρμόσουν αυτά τα οποία μαθαίνουν στο σχολείο στο λεγόμενο πραγματικό κόσμο μέσω διαπολιτισμικής επικοινωνίας ή κοινωνέργων με τους ε, ανθρώπους ίδια ηλικία από άλλες χώρες. Γι' αυτό πρέπει να συνεχιστεί μετά το 2020. Η Εστονία και άλλες χώρες θέλουν να υπάρξει ένα κεφάλαιο για την νεολαία με ξεχωριστό προϋπολογισμό. Αν δεν γίνει αυτό θα κινδυνεύσει η δουλειά που γίνεται στην νεολαία ως μια εκπαιδευτική προσέγγιση που έχει την δική του δική της αξία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επενθυμίζω ότι εμείς αγωνιστήκαμε στο Κοινοβούλιο για να υπάρχει ένα ποσοστό που να αποδίδεται σε επιμέρους προγράμματα. Αλέξανδρος Ζελτίνης από τη Λιθουανία. Ευχαριστώ. Ε, εξ ονόματος της, ε, του Λιθουανικού Κοινοβουλίου θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτή την ε, συνεδρίαση που είναι πραγματικά κρίσιμη. Η διαβίω εκπαίδευση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της εθνικής, ε, ε, του Εθνικού Προγράμματος της Λιθουανίας 2013-2022. Ε, θέλουμε, μάλλον θέσαμε το 2014 την μείωση της ανεργίας των νέων ως βασικό μας, βασική μας προτεραιότητα. Η Λιθουανία μάλιστα έχει σημειώσει πρόοδο σε ό,τι αφορά τους ε, στόχους ε, του, για την εκπαίδευση ε, στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρώπη 2020. Η απόκτηση του διπλώματος και η μείωση της σχολικής εγκατάλειψης συγκεκριμένα είναι δείκτες στους οποίους έχουμε βελτιωθεί πολύ. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όμως τα προβλήματα της αναντιστοιχίας ε, των δεξιοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διαβίου μάθηση και να επιταχύνουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση. Όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε μέσω της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στους ε, νέους ε, ανέργους ε, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης. Στην Ευρώπη η άτυπη εκπαίδευση γίνεται όλο και πιο σημαντική. Θέλουμε να σας υπογραμμίσουμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για την νεότητα θα πρέπει να καλύπτει όλους τους νέους. Όλους τους νέους που επιθυμούν να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς που έχουν φιλοδοξίες. Ευχαριστώ. Κύριε Βράιεν. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Ο προπολογισμό ε, για το Erasmus Plus έχει αυξηθεί κατά 40% αλλά ε, τα πρώτα χρόνια δεν φαίνεται αυτό. Ε, αυτό το οποίο έχει επικριθεί είναι ότι κάποια συγκεκριμένα προγράμματα όπως το Comenius μέσω της αναδιάρθρωσης των προγραμμάτων διαθέτουν λιγότερα λεφτά απευθείας ε, στα σχολεία και στις σχολές ε, και ανταυτού πηγαίνουν σε κάποια έργα τα οποία βεβαίως ε, αφορούν την συνεργασία των σχολείων. Και ίσως γίνεται κάποια κατάχρηση του Εράσμους καθώς μειώνονται τα κονδύλια για το Horizon 2020 κτλ. Και ε, δεν ξέρω, το βλέπετε και εσείς αυτό ότι μπαίνουν ε, κάποια στιγμή τα πανεπιστήμια και παίρνουν τα λεφτά τα οποία προορίζονταν ίσως για σχολεία κτλ. Σας ευχαριστώ, Birgit Young. Ο κύριος Young έχει το λόγο και μετά ο Ιπνιρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να πω είναι το κατά πόσον ε, τα προγράμματα αυτά απευθύνονται στους νέους ε, που πραγματικά τα χρειάζονται. Η εμπειρία μου από την Αυστρία είναι πως ε, τα προγράμματα αυτά τα χρησιμοποιούν αυτοί οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν το επίπεδο για να τα εκτιμήσουν. Και δεν βλέπω τα προγράμματα αυτά να εφαρμόζονται εκεί όπου υπάρχει ίσως μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί όπου δεν υπάρχει και τόση γνώση. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι ίσως κάπως πιο στοχευμένα. Σας ευχαριστώ. Ευντυρό από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στη Γαλλία Έχουμε ισχύσει ένα σύστημα για τι απαντήσει των 150.000 νέων που εξέρχονται του συστήματος ε, δηλαδή όχι μόνο από τα σχολεία αλλά και από την ιδιότητα του πολίτη, την ηθαγένεια. Τώρα, πώς μπορεί λοιπόν αυτό να ε, συμπεριληφθεί στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών πρώτο ερώτημα και σε ό,τι φορά την αγωγή του πολίτη και τα δεξιότητε που έχουν αποκτήσει μπορούν να ε, συμπεριληφθούν σε ένα είδος ευρωπαϊκού διπλώματο. Ευχαριστώ, θα απαντήσω θα απαντήσουμε μετά. Μετά το λόγο έχει η κυρία Ward. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι Είμαι από του συνάδελφου που έφτασαν αργότερα στην αίθουσα διότι ήμουν στη συνεδρίαση των Επιτροπή Γυναικών που ασχολούνται με την φτώχεια, με την ένδια. Η ένδια δεν είναι κάτι μόνο το υλικό, αλλά είναι και ένδια ευκαιριών. Θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφος μιλούσε για την επιστροφή στα σχολεία των νέων Έχουμε στην πατρίδα μου κάποια προγράμματα τα οποία βασίζονται σε εξετάσεις ε, και είναι πολύ τυποποιημένη η παιδεία και δεν ε, έρχονται συχνά σε επαφή με άλλες, ε, άλλους πολιτισμούς. Θα ήθελα να πω ότι στους όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τους ε, μαθητές αλλά και τους καθηγητές, τους δασκάλους και ούτω καθεξής. Και αυτά οι άνθρωποι χρειάζεται να γνωρίζουν γιατί είναι τόσο σημαντικό να ε, βγαίνουν έξω από τα σύνορα της χώρας τους διότι όταν συμβεί κάτι τέτοιο μπορεί να αλλάξετε άρδιν αλλά γίνεται άλλος, άλλος άνθρωπος αν γνωρίζετε άλλους πολιτισμούς και άλλα κράτη και να μην πτωχεύουν μόνο σε εξετάσεις και στους ε, σημαίνει στόχους. Ο κύριος ε, Βουλκάνης, πρόεδρος της Επιτροπής στην Εθνικό του Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Μιλώ εκ μέρους της αντιπροσωπής της Λετωνίας και θα ήθελα να σας μιλήσω για τη δική μας εμπειρία σχεδιασμού της ε, πολιτικής νεολαίας. Εμείς δημιουργήσαμε το Κοινοβούλιο των Νέων στην Λετωνία και είναι ένας ε, θεσμός ο οποίος ε, προσπαθεί να κατανοήσει τον τρόπο λήψη αποφάσεων μια δημοκρατική κοινωνία και να το βελτιώσει. Δεύτερον, η... στη Λετωνία δρόνωσα μια συζήτηση στο κοινοβούλιο μας για την, ε, περίπτωση μείωσης του ορίου ε, ε, για την απόκτηση του δικαιώματος ε, να ψηφίζουν οι νέοι από τα 16 ακόμα δεν υιοθετήθηκε όμως αυτό το μέτρο. Έχουμε κάνει πολλά για να διεθνοποιήσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Διαθέτουμε νομοθεσία που μας δίνει τη δυνατότητα να διοργανώνουμε κοινά προγράμματα, ε, εκπαιδευτικά προγράμματα με σχολεία και πανεπιστήμια άλλων χωρών, καθώς επίσης ε, και με τεχνικές σχολές και ε, σχολεία κατάρτισης. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα πρόταση. Γνωρίζω πως κάποια κράτη έχουν ιδρύσει ή περιφερειακά τοπικά κοινοβούλια με ή να έρθουν σε επαφή με τους νέους για να απαντήσει τώρα θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν νομίζω ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες διευκρινείς που μπορούν να μας δώσουν και οι δύο εισηγητέ από δύο λεπτά μέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά διότι θα αναφερθώ σε πολλά ζητήματα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που καλέσατε και την Κομισιόν ε, και να ευχαριστήσω τον κύριο Λόπες για τα καλά νέα που μας έφερε για τους οργανισμούς που συμμετέχουν στην πλατφόρμα για την διαβίου κατάρτιση και βλέπουμε πως πάνω από το 80% είναι ικανοποιημένοι με το πως ε, ανταποκρίνεται το πρόγραμμα Erasmus Plus στους στόχους που έχουν τεθεί και στις ανάγκες ε, των δικαιούχων. Ε, θα ήθελα να τονίσω πρώτα απ' όλα πως τα αποτελέσματα των πρώτων δύο ετών ε, είναι αρκετά ικανοποιητικά. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ήδη αποφελήθηκαν από τις δυνατότητες κινητικότητας που μας δίνει το πρόγραμμα Erasmus Plus ε, το οποίο βέβαια κυρίως αφορά την κινητικότητα, αλλά ε, αναφέρθηκαν και οι άλλες πτυχέ. Ε, τα νέα τμήματα του Erasmus Plus, ειδικά αναφέρθηκε η διατομεακότητα και ε, τα νέα αυτά στοιχεία, ακριβώς επειδή είναι νέα, δεν είναι ακόμα τόσο επιτυχή όσο θα θέλαμε, οπότε, υπό μια έννοια, οι δικαιούχοι προηγούμενων προγραμμάτων και σε γενικές γραμμές οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε διάφορους ε, κλάδους δεν είναι μαθημένοι να δουλεύουν διατομεακά. Οπότε κατά κάποιον τρόπο δεν προξενεί εντύπωση το ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να μάθουν ακριβώς ε, το πρόγραμμα οι δικαιούχοι. Ταυτόχρονα βλέπουμε πως υπάρχει ενδιαφέρον. Ήδη το 2014 χρηματοδοτήσαμε σχεδόν 2.000 έργα. Για την ακρίβεια 1.700 ε, στρατηγικές ε, συνεργασίες. ...10.000 εκ των οποίων έχουν και διατομειακό ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα θα έλεγα πως ε, αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία στο να ανταποκριθούμε στο ενδιαφέρον που υπάρχει γιατί εκεί πέρα υπάρχει και το θέμα του υπερπολογισμού. Μέχρι στιγμή, βεβαίω έχουμε όπω είπαμε ένα ποσοστό επιτυχία 18% αλλά αυτό οφείλεται στον ε, προπολογισμό. Τα επόμενα έτη θα έχουμε μια αύξηση κατά 80% του προπολογισμού μέχρι το 2020 και αύξηση 50% για στρατηγικέ συνεργασίε και διατομιακέ. Ε, δραστηριότητες. Επίσης, οι περιορισμοί αυτοί του προπολογισμού ισχύουν και για την δράση κλειδί, όπως λέμε, την υπαριθμόν 3, που αφορά δραστηριότητες που κοιτάνε περισσότερο τον διάλογο και τον πειραματισμό για ζητήματα χάραξης πολιτικής και εδώ πέρα ακριβώς σκοπεύουμε να αυξηθεί και αυτός ο προπολογισμός όταν αυξηθεί ο γενικότερος προπολογισμός. Γι' αυτό, ε, ναι, τελειώνω. Γι' αυτό είναι σημαντική αύξηση του προπολογισμού και διαβεβαιώ του ε, βουλευτές, ε, τους και τι βουλευτές που ασχολούνται ε, και με το θέμα της ανώτατη εκπαίδευση σε σχέση με τους άλλους κλάδους. Θα σεβαστούμε τα ποσοστά που αναφέρονται στην νομική βάση για το κάθε κομμάτι και ταυτόχρονα να τονίσω πως ε, έχουμε μια στρατηγική ακριβώς για να ευνοήσουμε μειονεκτικές ομάδες και βλέπουμε πως 30% ε, των δικαιούχων είναι από αυτές τις ομάδες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι διευκρινήσεις για τον προπολογισμό. Ελπίζω του χρόνου να υπάρξει αυτός, αυτή η αύξηση. Είχαμε ένα πρόβλημα ειδικά με τις πληρωμές ε, που προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε δεσμεύσαμε 6 εκατομμύρια πλέον για το Εράσμος. Ε, πραγματικά δύο λεπτά έκαστος. Σύντομα για δύο λεπτά πρόεδρε. Πρώτον, ένα ουσιαστικό ζήτημα είναι η σύνδεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να στηρίξουμε τα διαβήματα προς τα κράτη. Οι παρεμβάσεις τόσο των Ευρωβουλευτών όπως η κυρία Τζούλιο, ο κύριο Νίκοφ ε, ή ε, ακόμα και οι εθνικοί βουλευτές που μίλησαν κατέληξαν ότι είναι απαραίτητος, απαραίτητο διότι ε, ο προπολογισμό εξαρτάται από τα οράματα των κράτων μελών. Δόθηκαν πολλά χρήματα για την κατασκευή δρόμων, οδών, αλλά βρούμε σήμερα χρήματα για την εκπαίδευση. Πρέπει να ενισχύσουμε τον διάλογο ανάμεσα στην κοινωνία και τα θεσμικά όργανα. Έχουμε ένα πολύ καλό εργαλείο, το άρθρο 11 της Συνδίκης Λισαβόνας, που βασιστούμε σε θετικότατες ε, εμπειρίες ηλιοσύλλα ε, από τον ε, φόρουμ της νεολαίτητας αναφέρθηκε. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε στο σύνολο της κοινωνίας των πολιτών, στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, για να ξεφύγουμε από το πλαίσιο του στενού λόμπι. Ευχαριστώ τηλεγραφικός ήσασταν. Όταν ε, μιλάω λοιπόν για το τι κάνουμε, ένα από τα πράγματα τα οποία ανέκαθεν θίγω είναι ότι οι ανταλλαγές είναι ιδιαίτερα ελιτιστικές. Γι' αυτό και ένα κομμάτι του πληθυσμού δεν συμμετέχει. Να τονίσω ότι δεν πρέπει να δούμε αυτές τις ανταλλαγές ώστε να δώσουμε απλά πλέον εκτίματα σε κάποια πρόσωπα. Αυτές οι ανταλλαγές, δόξα τω Θεώ, είναι ένα καλοπτικό σύστημα, είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε, διότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι ε, το θεμέλιο του συντηρητισμού και του εθνικισμού. Να το αναγκάσουμε τα σχολεία να έρχονται σε επαφή με σχολεία άλλων χωρών και να ανταλλάσσουν μαθητές φοιτητές είναι καλύτερη διαδικασία. Το 50% των ευρωπαϊκών χωρών δεν δίνουν καμία αξία στο να πάει ένας μαθητής ή ένας φοιτητής στο εξωτερικό για ένα χρόνο διότι όταν πηγαίνει σε άλλο κράτο θεωρούν ότι δεν μαθαίνει τίποτα. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και να το βελτιώσουμε. Η μεγαλύτερη επένδυση λοιπόν θα πρέπει να γίνει από πλευρά κομισιών στο να διεθνοποιεί, τα, διεθνοποιήσει τα εθνικά μας συστήματα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει ένας πραγματικός διάλογος ανάμεσα σε ισότιμους αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητό. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειε δεν πάρει το χρόνο, αλλά το 60% ε, των, ε, ε, των, φοιτητών στην Ιταλία δεν έχουν μεταβεί στο εξωτερικό, δεν μιλάνε ξένη γλώσσα, δεν έχουν σε επαφή με ξένους, με αλλοδαπούς. Κανείς λοιπόν δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με, το, με εκπαιδευτικά προγράμματα και θέματα διδασκαλίας αν δεν έχει ε, ζήσει και στο εξωτερικό, αν δεν έχει εκπαιδευτεί και στο εξωτερικό. Είναι κάτι σκέψη, θα το σκεφτούμε. Να υπενθυμίσω πως ε, εμείς τα προγράμματά μας ε, βγάλαμε ότι μέχρι το 2020 ένα σημαντικό ποσοστό, δεν θέλω να πω κάποιο ποσοστό λάθος, νομίζω 20% είναι ήδη ένα μεγάλο ποσοστό διότι το Erasmus ε, τώρα θα αφορά για τα 7 πρώτα χρόνια τα 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν στους στόχους μας ε, θέσαμε τουλάχιστον 20% των παιδιών θα πρέπει να έχουν κάνει όχι μόνο το εράσμος αλλά και μια περίοδο κατάρτισης, επιμόρφωσης σε άλλο κράτος. Για μας λοιπόν το θέμα είναι κεντρική σημασίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτό το σημαντικό πάνελ που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Θα συνεχίσουμε την επαφή μας, δεν θα χαθούμε. θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ, ε, διαπολιτισμικός διάλογος μέσω της ε, εκπαίδευση. Έχουμε δύο συμμετέχοντες στο πάνελ ε, με διαφορετικές προσεγγίσεις, θα ακούσετε το γιατί. Πρόκειται για τον Μεσημιλιάνο Μοσκερίνη για την για την κοινωνική ένταξη των νέων που είναι από την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την βελτίωση των ε, εργασιακών συνθήκων και μετά θα δείτε και ένα πολύ ωραίο φιλμ για τον διαπολιτισμικό διάλογο ο καθηγητής Μασκερίνη παρακαλώ να λάβει το λόγο ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Από την οπτική γωνία ενός νέου κοινωνική ένταξη μπορεί να ειδωθεί ως η πραγμάτωση του δυναμικού του νέου στην κοινωνία και ταυτόχρονα αναγνώριση από πλευρά της κοινωνίας αυτού του δυναμικού και αυτό μπορεί να γίνει μέσω τριών τρόπων κυρίως ε, ε, εκπαίδευση, εθελοντισμός και κοινωνική συμμετοχή καθώς επίσης και απασχόληση. Ε, η έννοια της κοινωνικής ένταξης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους, αυτούς που, έχουν τα, που βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση. Όπως είπα και πριν, οι νέοι είναι αυτοί που πιο πολύ υφίσταν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη σήμερα. Η κατάσταση έχει χειροτερεύσει αρκετά σε σχέση με το 2008. Σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από το 1 τέταρτο των νέων αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ε, ιδιαίτερα οι νέοι που είναι εκτός εργασίας, εκτός εκπαιδευτικού συστήματος ε, και εκτός κατάρτισης. 14 εκατομμύρια ε, άτομα στην Ευρώπη, κάτω των 30, ε, βρίσκονται, σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή. Με ένα, ε, με ένα τεράστιο κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ενσωματώσουμε τους νέους στην αγορά εργασία και να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, ε, το House μάλλον το Κοινοβούλιο ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νεολαία του 2010 9 έτσι ώστε να δώσουν με στους νέους ίσες ευκαιρίες στην ε, εκπαίδευση και στην αγορά και να ενθαρρύνουμε τους νέους να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες στην κοινωνία μας. Η εφαρμογή της στρατηγικής για την νεολαία έγινε με δύο πυλώνες. Πρώτον η απασχόληση που είναι ε, που εισιτήριο για πολλές δραστηριότητες και μια πιο ευρεία αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ε, σε ό,τι αφορά την απασχόληση μέσω της, συστήματο ε, συστήματος εγγύησης για την νεολαία, ενώ ε, σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα με διάφορες υπηρεσίες, συμμετοχή και ειδική βοήθεια για τις μειονεκτούσες ομάδες. Σε ό,τι αφορά την εγγύηση για την νεολαία, ε, δίνει την ευκαιρία για απασχόληση, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία και κατάρτιση ε, σε περίοδο τεσσάρων μηνών από την στιγμή που κάποιος χάνει τη δουλειά του ε, ή φεύγει από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκπαίδευση είναι το πρώτο σημείο εισόδου της κοινωνικής ένταξης και δίνει τη δυνατότητα στους ε, νέους να μπουν στην, Ευρωπα... στην αγορά εργασίας αλλά και να γίνουν και πολίτες. Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου είναι η... Ε, ε βασικός παράγον είναι η πρόορη εγκατάλειψη του εκπαιδευτικού συστήματος. Ε, αυτοί έχουν τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αποκλειστούν. Ένα από του βασικούς στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι αυτός να καταπολεμηθεί η πρόορη εγκατάλειψη σχολείου. Ε, η σε φορά την εκπαίδευση έχουμε ε, μια προληπτική προσέγγιση με πολιτικές ε, γεωγραφικά προσδιορισμένες αλλά και ταυτόχρονα με τη δημιουργία εναλλακτικών περιβαλλόντων μάθησης με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας με παροχή συμβουλών και προσανατολισμού. Εδώ έχουμε ε, και δεύτερον έχουμε το δεύτερο πυλώνα της επανένταξης με διάφορα παραδείγματα όπως η κοινότητα αν, μάθησης της Ισπανίας αλλά και ε, ε, τα μαθήματα Mosaic στο Λουξεμβούργο που είναι εναλλακτικέ μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί. Μετά, Έχουμε ε, σε ό,τι αφορά την επανένταξη έχουμε εναλλακτικέ ε, μεθόδους ε, σε μια πιο επίσημη βάση, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γλωσσικά μαθήματα για τους μετανάστες, αλλά και αντιμετωπίζουν και πιο περίπλοκες ανάγκες, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα των σχολείων της γειτονιά στην Ολλανδία, που προσπαθεί να καλύπτει τις ανάγκες ιδιαίτερων ομάδων του πληθυσμού που δεν μπορεί να τις καλύψει η επίσημη εκπαίδευση. Στην Γαλλία ονομάζονται σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Ε, ως συμπέρασμα χρειαζόμαστε περισσότερη ε, σημασία να δώσουμε στην κοινωνική, στον κοινωνικό αποκλεισμό των νέων και κάτι το οποίο πηγαίνει πέρα από το θέμα της ε, ανεργίας. Ε, τα κράτη-μέλη άρχισαν να εφαρμόζουν το σύστημα της ε, εγγύησης νεολαίας. Ε, είναι ένα εργαλείο για την στρατηγική για την νεολαία του 2009. Η εκπαίδευση έχει να παίξει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εγγύηση για την νεότητα. Είναι το πρώτο σημείο εισόδου για τις πολιτικές κοινωνικού ένταξης για τους νέους και θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης που θα συμπεριλαμβάνει και την εκπαίδευση και την απασχόληση αλλά και μια πιο ευρία αντιμετώπιση της κοινωνικής ένταξης ιδιαίτερα για τους πιο μειονεκτούντες όπως οι πρόσφυγες κλπ. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω αν ε, κάποιος θέλει να λάβει το λόγο. Α, ένας έχει ζητήσει το λόγο. Πρώτα έχουμε το European Youth Forum. Συγγνώμη, συγγνώμη, λάθος. Μάλλον η κούραση. Τα φταίει. Το λόγο έχει η δεύτερη κυρία του πάνελ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για το πρόγραμμά σας, ο κυρία Σέρνερ και μετά το Youth Forum. Möjligheten att få komma hit och berätta om er Det är med stor Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω να σας μιλήσω για το τι κάνουμε στην Σουηδία και σε άλλες ευρωπαϊκές ε, χώρες. Το Μάιο του 2009 ένα σχολείο στο Γκέτεμπορκ δέχτηκε μία προσφορά από το Υπουργείο Παιδείας ε, να πάνε σε ένα γυμναστήριο να ακούσουν ε, κλασική μουσική από ζωντανή ορχήστρα και ήταν πάρα πολύ φορά πολλοί από εμάς άκουσαν Μπετόβεν κτλ και θα ήθελα να πω πως η μουσική ε, το συζητήσαμε στην Άλφο και με ρώτησε αν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο ειδικά για τα παιδιά και λέει πως μπορούμε πράγματι να το χρησιμοποιήσουμε και έτσι όντως έγινε μετά έλαβε και ένα βραβείο στην Βενεζουέλα ε, για το ότι έδωσε χιλιάδες παιδιά την ε, ευκαιρία να ξεφύγουν από τη φτώχεια με την ε, μουσική και έδωξε, έδειξε επίσης πως η μουσική μπορεί να γεφυρώσει τα χάσματα και να μπορέσει να φέρει κοντά ανθρώπους σε μια διαχωρισμένη πόλη όπως το Γκέτεμποργκ. Έχουμε κόσμο που ζει χωριστά, ανθρώπους που ζουν σε δύσκολες συνθήκες και έχουμε ακριβώς αυτά τα μουσικά και πολιτισμικά σχολεία. Κάναμε μάθημα μουσικής σε πάρα πολλά παιδιά και σιγά σιγά τώρα έρχονται και άλλα παιδιά και έχουμε μία νέα πρόκληση στο πολιτισμικό αυτό σχολείο και έτσι μπορούν τα παιδιά να δουν πόσο συναρπαστική μπορεί να είναι η μουσική έτσι έχει δημιουργηθεί ένα σουηδικό μοντέλο όπου η μουσική συνεισφέρει στην ε, κοινωνική ένταξη. Και επίσης έχουμε μουσικούς οι οποίοι πηγαίνουν στα σχολεία, συναντάν τα παιδιά και είναι μετά πάρα πολύ σημαντική η δυνατότητα. Τα παιδιά παίζουν για τους γονείς τους, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επαφές. Ε, υπάρχουν λοιπόν αυτές ε, οι πολύ σημαντικές επαφές και ανάπτυξη και των γλωσσικών δεξιοτήτων. Λοιπόν, το ελσιστέμα στην Σουηδία δραστηριοποιείται σε 20 δήμους ε, γύρω στα 7.000 ε, παιδιά ε, έχουν περάσει από το πρόγραμμα και έτσι νομίζω πως ε, μπορούμε να φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά. Έχει διαδοθεί το σύστημα ε, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οργάνωση πλέον ε, σε Αυστρία και Μεγάλη Βρετανία και δραστηριοποιούμαστε όπως σας είπα σε διάφορες ε, χώρες και και στη σκάλα του Μιλάνου είχαμε συναντηθεί, κάνουμε διεθνείς συναντήσεις συχνά έρχονται νέοι σε επαφή, μαθαίνουν για την ε, μουσική και στο ραμπλόχ στην Σκοτία επίσης ε, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και δίνονται νέες δυνατότητες στους παιδαγωγούς ε. σε 65 χώρες λοιπόν υπάρχει το σύστημα είναι πάρα πολύ διαδεδομένο δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος, απλά το μήνυμα από την Βενεζουέλα είναι ότι πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί αυτόνομα. Και βλέπουμε πως έχουμε ανά τον κόσμο ένα εκατομμύριο παιδιά που ασχολούνται πλέον με την μουσική από μικρά, κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει σε όλη την ζωή τους ε, και ελπίζουμε έτσι να αποφύγουν την εγκληματικότητα και τους ε, δρόμους. Παραδείγματος χάρη είχαμε και ένα κοριτσάκι που είχε μια αλκοολική μητέρα και τελικά κατάφερε σε αυτού του προγράμματος και η μητέρα της να βρει φίλες και η σχέση μητέρας και κόρης αναπτύχθηκε και μας είπε πως μέσω του συστήμα ξανακέρδισε τη μητέρα μου. Η Αντέλα από το Ιράκ βρίσκει εκεί πέρα διέξοδο από τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι της ε, και η Μίκε είχε έρθει από την Χιλή πριν από μερικά χρόνια μέσω του συστήμα γνώρισε την Σουηδία και προσκλήθηκε και η οικογένειά της σε διάφορα, διάφορες συναυλίες αυτά και υπάρχουν οπωσδήποτε και άλλες ε, περιπτώσεις ε, λοιπόν υπάρχει πολύ έντονη δραστηριότητα στο Γκέτεμποργκ και βλέπουμε πως η μουσική γεφυρώνει τις ε, διαφορές ε, των ανθρώπων ε, και δημιουργεί πράγματι ένα κλίμα συνεργασίας και πειθαρχίας πράγματα που χρειάζονται στην ε, καθημερινή ζωή, επαφή με άλλους ανθρώπους, με άλλα επαγγέλματα και έτσι γίνονται τα παιδιά καλύτεροι πολίτες. Λοιπόν, έχουμε ένα βίντεο κλιπ ε, το οποίο θα σας ε, δείξουμε τώρα στις οθόνες πόσο 20 δευτερόλεπτα tengan acceso a, la, a, a, a más puro,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 Ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, δεν χρειάζονται σχόλια για το πως ε, η μουσική μπορεί να είναι ένα σύστημα ένταξης ε, αλλά και επιστροφής στην τυπική εκπαίδευση. Ίσως θα μπορούσαμε να ανάψουμε τα φώτα τώρα. Είπατε πως Ανοίγω παρένθεση, εγώ θυμόμουν τον ε, Χωσέ Εμπρέου που εφήβριε αυτό το σύστημα στην ε, χώρα του και τώρα έχει μεταφερθεί και στην Σουηδία. Να υπενθυμίσω λοιπόν πως αυτό το σύστημα εφαρμόζεται σε διάφορα κράτη τώρα. Να πω επίση ότι στην Ιταλία ε, θα γίνει ένα κοντσέρτο στην Γερουσία στις 20 Δεκεμβρίου. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο των νέων. Young Wilker, το Youth Forum και μετά θα λάβουμε το λόγο δύο συνάδελφοι και θα περάσουμε μετά στο τρίτο πάνελ. Ευχαριστώ. Το European Youth με τα χαρά συμμετέχει σε αυτό το ζήτημα. Όπως ε, τονίσαμε είναι νέοι πλήγησαν σκληρότερα από την κρίση και ακόμα υποφέρουν. Δυστυχώς η συζήτηση στα ΜΜΕ έχει ασχοληθεί περισσότερο με τον εξτρεμισμό, τη βία και ακόμα και την τρομοκρατία, αλλά εμείς θεωρούμε πως οι νέοι πρέπει να έχουν μια φωνή σε αυτή τη συζήτηση για διατομεακά προγράμματα με άλλους ε, κλάδους για να προωθήσουμε ακριβώς τα ζητήματα της ένταξης διαπολιτισμικού διαλόγου όπως αυτό το l παραδείγματος χάρη θεωρούμε πως αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να τα διδάξει κανείς πρέπει να τα ζήσει ε, και να υπάρχουν ακριβώς ε, κάποια ασφαλείς χώροι εντός των κοινοτήτων και συχνά η κινητικότητα των νέων περιορίζεται λόγω ακριβώς των δυνατοτήτων που δεν έχουν οι ε, για να μπορούν να κινούνται στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που θίξατε αυτό το ζήτημα. Δώσω το λόγο στους τέσσερις εγγεγραμμένους, Φιλίπ Λέξφελντ από την Γερμανική Βουλή. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δουλευτής Βερολίνου είμαι. Θα ε, ήθελα να πω κάποια πράγματα. Έχω μία ερώτηση για αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Μασκερίνη. Ε, στους στόχους ε, συμφωνούμε, αλλά έχω την εντύπωση πως η εικόνα είναι κάπως μονόπλευρη δεν ξέρω, ίσως έχω επηρεαστεί από το Βερολίνο. Τι γίνεται με το θέμα της αποδοχής των ευρωπαϊκών αξιών της δημοκρατίας, της ισότητας των γυναικών, του δικαιώματος ε, του Ισραήλ να υπάρχει. Όλα αυτά παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο και δεν τα άκουσα από εσάς. Ε, dopo diamo la parola ai nostri interlocutori e prima dare la parola a Yanis Vukanis di eh, Latvia. Yanis Vukanis από τη Λετωνία. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξαναπάρω το λόγο. Συμφωνώ με τον Μασιμιλιάνο Μασερίνη για ανεπαρκής εκπαίδευση αποτελεί αιτία κοινωνικού αποκλεισμού. Εγώ θα έλεγα κοινωνικής απομόνωσης από την κοινωνία. Η Λετωνία είναι μεταξύ των χωρών που άρχισαν να εφαρμόζουν το σύστημα της έγκυσης για την νεολαία αλλά αυτό αντιμετωπίζει τι συνέπειε όχι τι αιτίε. Για να αντιμετωπίσουμε τις αιτίε χρειαζόμαστε προληπτικά μέτρα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να βελτιωθεί η επαγγελματική κατάρτιση. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναπτύξουμε το σύστημα της διτής εκπαίδευση, μαθητεία και κατάρτισης. Η ιδέα μας είναι να ε, πείσουμε και να, να, να επιτρέψουμε στους εργοδότες να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό. Και έχουμε στρατηγική γι' αυτό. Προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει... Συγγνώμη. Η κυρία Σάνα Λαουσλάντη από τη Φιλανδία. Και μετά εσείς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στην Φιλανδία θεωρούμε ότι το σύστημα εγγύηση στην νεολαία είναι εξαιρετική ιδέα. Θα έχουμε, το έχουμε ξεκινήσει αλλά πρέπει να το βελτιώσουμε και να το αναπτύξουμε περαιτέρω. Χρειαζόμαστε δράση πριν ξεκινήσουν τα παιδιά το σχολείο. Οπότε πρέπει να δούμε τι δεξιότητες χρειάζονται πριν ακόμα ξεκινήσουν τη σχολική τους εκπαίδευση. Εμείς έχουμε μετανάστες, γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι η γλώσσα χρειάζεται πριν ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους. Χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε τις γλωσσικέ τους δεξιότητες πριν από τη σχολική του ηλικία. Και αυτό το λόγο έχουμε ένα συστητικό σύστημα τριών επιπέδων. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε όλους τους μαθητές στο σχολείο έτσι ώστε να μην έχουμε πρόορες εγκαταλείψεις. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να δράσουμε πριν ξεκινούν στο σχολείο και ε, θα πρέπει να αναπτύξουμε τέτοιου είδου ε, συστήματα. Του χρόνου θα πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. E Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα. Ο κύριος Βέντα. Πώς μπορείτε να ζητήσετε λόγο στον επόμενο γύρο. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Ο κύριος ο είπε ότι ο αθλητισμός είναι η κοινή γλώσσα κατανοητή, αλλά και η μουσική και η γλυπτική είναι ιδιαίτερα κατανοητές γλώσσες όπως και είναι εκπαιδευτικές μέθοδοι το σύστημα έχει κάποιες νέες μεθόδους. Είδα ότι υπάρχουν έλεγχοι, εξετάσεις. Μπορείτε όμως να μου πείτε πού βρίσκεται το σχετικό κέντρο για την Τσεχία. Ε, και αναφέρομαι στα όσα είπε στην στην Σουηδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα ο χρόνος ε, είναι πάρα πολύ φορτωμένος, πιεσμένος. Ε, η Επιτροπή μας οργάνωσε μια συνεδρίαση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Άκουσα διάφορα μέτρα για την κοινωνική ένταξη. Φυσικά μιλάμε για τους νέους, για τα παιδιά, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα άτομα, τα μερικές ανάγκες, τους αναπήρους. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία, μιλήσαμε για τη μουσική, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό. Εμείς χρησιμοποίησαμε την ε, μαγειρική για νέους ε, ε, οι οποίοι δεν έχουν πολλές δυνατότητες αλλά μπορούν να συμμετέχουν σε, για την προετοιμασία φαγητών, γευμάτων στην χώρα, στην πόλη μου. Έχει ανοίξει ένα ιδιαίτερα σημαντικό εστιατόριο για τους ε, κοφάλαλους. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές ε, για τη συνεργασία δύο κόσμων των ε, νέων που είναι υγιέστατοι και άλλων οι οποίοι είναι υγιείς αλλά έχουν κάποιο μειονεκτήματα. και το να μεταβαίνουμε, να πέφτει τα μετάβαση σε αυτά τα εστιατόρια είναι καλό διότι έτσι μπορούμε να δούμε πώς μπορούν να συνεχθούν τα πρόσωπα αυτά μεταξύ τους. Ευχαριστώ. θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπάρξει ε, μια περίληψη όλων όσων συζητώνται σήμερα, όλων των εμπεριών που ακούσαμε. Θα δώσω το, το λόγο στους ε, πανελίστες προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Λοιπόν, νομίζω πως Όπως ε, είπε και το Φόρουμ της Νεολαίας, η διατομιακή προσέγγιση είναι σημαντική όταν μιλάμε για τα ζητήματα των νέων, απασχόληση, ένταξη και εκπαίδευση. Γιατί όταν μιλάμε για την νεολαία, μιλάμε για έναν ολόκληρο γαλαξίο και μια διαφοροποιημένη προσέγγιση που είναι κομμάτι της εγγύησης για την νεολαία είναι πιο αποτελεσματική. Δεν γίνεται να κάνουμε τα ίδια για όλους, να μιλάμε για την ε, νεολαία, γιατί βεβαίως διαφέρει και το επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και κάποιες προσεγγίσεις μπορεί να λειτουργούν για κάποιους, όπως η μουσική παραδείγματο χάρη, ενώ άλλες, όπως ο αθλητισμός, για μια άλλη ομάδα νέων. Οπότε αυτός ο συνδυασμός ε, συνεργασίας μεταξύ διαφόρων θεσμικών οργάνων και κλάδων και η διαφοροποιημένη προσέγγιση και η ενεργοποίηση και η ένταξη των νέων σε εθελοντικές δραστηριότητες παραδείγματος χάρη ε, είναι το κλειδί της αποτελεσματικότητας της εγγύησης για την νεολαία που είναι ένα σημαντικό εργαλείο παρά το ότι σε κάποιες χώρες αυτά θα είναι πραγματική επανάσταση στην πολιτική για την νεολαία, αλλά είναι σημεία κλειδιά όπως ε, είπαν ε, και κάποιοι ομιλητές. Και από αυτό το πρίσμα η εκπαίδευση όπως είπαμε είναι ο τρόπος όχι μόνο να αποκτήσουν οι νέοι δεξιότητες για την αγορά εργασίας, αλλά να καταστούν ε, πλήρως ε, πολίτες της ε, κοινωνίας μας. Να αντιληφθούν και να μοιραστούν τις αξίες μας. Και όσον αφορά την αποδοχή των ευρωπαϊκών αξιών, όπως τονίσατε, νομίζω πως η ένταξη των ε, νέων ε, στην εκπαίδευση νομίζω θα είναι αποτελεσματικότερος τρόπος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω πως ε, σήμερα ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ήθελα να γνωρίζω, ίσως έχουμε και ευκαιρία να το συζητήσουμε και σε μεταγενέστερο στάδιο, η προσέγγιση σχετικά με την εγγύηση προς τους νέους θα πρέπει να είναι πιο ολιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή η ένταξη δεν είναι μόνο θέμα απασχόλησης, είναι ζήτημα ευκαιριών που δίνονται ολοκληρωμένες για την απόκτηση της, κατα... της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, αλλά και το στάζ, το πρόγραμμα σχετικά με τις ευκαιρίες των δυνατοτήτων, των ευκαιριών που προσφέρονται κάτι που σε περίοδο κρίσης ε, να μην είναι εύκολο εξέβρεση εργασίας αλλά υπάρχει και ε, πολιτική εμπειρία ή και ε, ανεξάρτητη θα μπορούσαν λοιπόν να υπάρξουν εργαστήρια, τα λεγόμενα hub αλλά και μια σειρά από άλλες ευκαιρίες, όχι παράλληλες, αλλά που ολοκληρώνονται στις διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση και σε επίπεδο ε, εθνικών και, και ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Δεν ξέρω αν στις χώρες σας, ε, στη δική μου τη χώρα, αλλά και εδώ, όλα αυτά είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και αρμόδιος είναι ο Επίτροπος ε, ζητήματα εργασίας. Αλλά το θέμα θα πρέπει να ειδωθεί ολιστικά. Θα ήθελα να γνωρίζω αν θέλετε να πείτε κάτι εσείς, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, θέλετε να πείτε κάτι, δεν νομίζω. Θέλετε, αν ναι, θέλω κάτι να σχολιάσω. Ε, ευχαριστώ. Να πω μόνο ότι το ελσιστέμα αναπτύσσεται στην Ευρώπη ε, λαμβάνει χρηματοδότηση και πολιτική στήριξη εργαζόμαστε σε μεγάλο βαθμό εθελοντικά θα σας θα στείλω τα στοιχεία στην ε, Τσεχική Δημοκρατία σε ό,τι αφορά τα μέτρα πρόληψης Είναι σημαντικό να εργαζόμαστε με τα παιδιά και για τα παιδιά πριν ξεκινήσει το σχολείο. Αυτό λόγο είναι σημαντική μουσική. Πριν ξεκινήσει το σχολείο. Ε, we'll any Πολύ ενδιαφέρον. Θα διανύμουμε οποιαδήποτε πληροφορίες μας στείλετε. Ανοίγω, ε, μάλλον, το, μάλλον ξεκινάμε. Το τελευταίο, τρίτο και πολύ σημαντικό πάνελ, δεν είναι πολιτικό πάνελ. Θα δώσουμε το λόγο σε τέσσερις εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων. Θα δώσω το λόγο στους εξβουλευτές Σάνα Σάβ Λάτε από τη Φιλανδία, Σαντρίν Ντουσέ από την Ελληνική Εθνοσυνέλευση. Αρχικά προβλέπεται ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης ε, της Ιταλικής Βουλής, Φραβία Ναρδέλη, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει σήμερα αλλά είναι η Φραντσέσκα Πουλίζη, η γερουσιαστής από την Ιταλία και Τζέρα Κραουβέλ, δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομα, από την Βουλή της Ιρλανδίας. Παρακαλώ, δύο λεπτά έκαστος. Ξεκινάμε με την Φιλανδία. Παρακαλώ. Το θέμα είναι η διαβίου μάθηση και η, ενεργός, και η ένταξη ενεργός ζωή. Ενώ προετοιμάζεστε να σας παρουσιάσω προσπαθούμε να έχουμε μία άποψη από τα διάφορα μέρη και περιοχές της Ευρώπης αλλά και από κράτη τα οποία έχουν ε, ε, μπλακεί πρόσφατα σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πλήρη μεταμόρφωση και είναι απολύτως ε, απαραίτητη ειδικά αυτή την εποχή γιατί στην αγορά εργασίας πολύ συχνά γίνεται αλλαγή εργασίας ε, παλιά κάποιο δούλευε στην ίδια θέση, στην ίδια εταιρεία για όλη τη ζωή, τώρα πια όχι. Αυτή τη στιγμή αλλάζουν ε, οι θέσεις ή ε, οι όροι εργασία, όπω για παράδειγμα μερική απασχόληση κλπ. Κάθε, όλο, γίνεται όλο και πιο δύσκολο κανείς να προετοιμαστεί για αυτήν την αγορά εργασίας. Οι συνθήκες αλλάζουν πολύ συχνά, είναι πολύ ρευστέ. Το μόνο σταθερό και σίγουρο είναι ότι αυτή η αλλαγή θα, είναι μόνο, θα, θα παραμείνει. Ε, αυτό, αυτή η καινούρια κατάσταση θα παραμείνει. Η, κατάσταση θα παραμείνει ρευστή γιατί ε, οι καινούριε τεχνολογίες, ε, η εισαγωγή των ρομπότ θα συνεχίζουν να ε, αλλάζουν το πανόραμα και τις δομές εργασίας. Θα γίνουν όλο και περισσότερη κατάρτιση εξ Αυτή τη στιγμή ήδη χρησιμοποιούνται πολλοί ρομπότ, θα χρησιμοποιούνται ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Ε, στις μεταφορές ενδεχομένως θα καταργηθούν ε, οι οδηγοί, στις μαζικές μεταφορές τουλάχιστον. Ε, ποια είναι η θέση της Ευρώπης και ποιες είναι οι δικές μας προοπτικές για το μέλλον. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε κατάρτιση διαβίου για να προσαρμοζόμαστε. Και αυτό αφορά όλους μας και όλες τις δεξιότητες. Στην Φιλανδία έχουμε αποφασίσει να αναμορφώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα επαγγελματική κατάρτισης, να το θέσουμε σε καινούρια θεμέλια, με καινούρια προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα, ε, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μέλλοντος. Θέλουμε να μπορούμε να δημιουργούμε και να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Και οι νέοι αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία χρειάζονται δεξιότητες, ικανότητες που να τους επιτρέψουν να μαθαίνουν καινούργια πράγματα, Καινούργι, να μαθαίνουν να, να, να μάθουν να μαθαίνουν. Και αυτό συνεχώς μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Γι' αυτό το λόγο η Φιλανδία ξεκίνησε από την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο μια δουλειά σε αυτό το θέμα και η οποία και συνεχίζεται. Ε, θέλουμε το, τα επόμενα χρόνια να αποτελέσουμε χώρα που θα είναι παράδειγμα σε ό,τι αφορά την διαβίου κατάρτιση και επιμόρφωση. Και θέλουμε αυτή να είναι προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες κάθε ανθρώπου. Επίσης, κατάρτιση από πιο νωρί και προσαρμοσμένη σε αυτό που θα χρειαστεί στο μέλλον. Οι καθηγητές μας θα πρέπει επίσης να επιμορφώνονται και να προετοιμάζονται πολύ καλύτερα για να αντιμετωπίσουν μαζί με τους μαθητές τους και τους φοιτητές τους αυτές τις προκλήσεις. Όλα έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση, προφανώς, και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από την ψηφιοποίηση και από τις ε, δυνατότητες που δίνονται ε, από την πληροφορική, έτσι ώστε τα συστήματα διαβίου κατάρτισης να είναι προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες, εξατομικευμένα. Ήδη ξεκινήσαμε με τα πρώτα βήματα. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα πανεπιστημίων και σχολών έτσι ώστε να είμαστε δημιουργικοί στο μέλλον και το εκπαιδευτικό σύστημα να στηρίζει αυτή τη δημιουργικότητα. Σε τοπικό επίπεδο έχουμε πλέον και παραδείγματα σε ό,τι αφορά τη, τόσο τη δευτεροβάθμια όσο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση με όλο και πιο στενούς δεσμούς με την αγορά εργασία και με τις επιχειρήσεις του χρόνου θα υλοποιήσουμε καινούρια εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια γιατί αυτά θα αποτελέσουν την στέρεη βάση που θα μας προετοιμάσει για το μέλλον. Θέλουμε να βελτιώσουμε το διάλογο καθώς επίσης και την κατάρτιση στα μαθηματικά και τις επιστήμες, θετικές επιστήμες και επίσης να προωθήσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα, την επιχειρηματική συνείδηση προκειμένου το μέλλον μας να είναι βιώσιμο. Γι' αυτό όμως χρειαζόμαστε και κοινωνική στήριξη. Θα πρέπει να μπορούμε να ακολουθήσουμε τη ροή της πραγματικότητας και να δώσουμε στους ανθρώπους μας τις κατάλληλες ικανότητες για να αντιμετωπίσουν το μέλλον. Με, ε, έχοντας ε, δει την έναρξη της, ε, ε της ψηφιακής επανάστασης θα πρέπει να προετοιμάσουμε την κοινωνία μας για μια νέα μεταμόρφωση, ένα καινούριο πολιτισμό και το εκπαιδευτικό ε, ε, σύστημα έχει να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να μιλήσουμε για το τι είναι το ταλέντο τόσο στην ε, εργασιακή ζωή όσο και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Αυτή ε, στην εποχή μας το στρες ε, είναι ένας βασικός εχθρός και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στην, ε, στις αλλαγές που στο σύστημά μας. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στα, στους εργαζόμενους και στους ε, νέους ε, να αναπτύσσουν το δυναμικό τους και εκεί οι επιχείρησεις έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Παρακαλώ να παραμείνετε στα δύο λεπτά προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτό το πάνελ και να δώσουμε ευκαιρία να λάβουν το λόγο και όσοι θελήσουν. Η Σαντρίν Ντουσέ έχει το λόγο που ακούσαμε και πριν από την μετροσυνέλευση της Γαλλίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μιλήσω ενώπιον σας ή να προσπαθήσω να σας παρουσιάσω ένα σύστημα πολύ περίπλοκο, το σύστημα ε, εκπαίδευση ε, ε, στη Γαλλία που είμαι λοιπόν μέλος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Επιτροπής εκπαίδευσης και παιδείας. Συμμετέχω και στα προγράμματα το 2013 και συμμετείχα στα σχολικά προγράμματα σχετικά με το πρόγραμμα που είναι κάτι το καινούριο στην Γαλλία όλων εφαρμόζεται εδώ και σε αρκετές χώρες ε, και βασιζόμαστε σε εμπειρίες που ιδιαίτερα επικοδομητικές. Εκλήθην για την ανάπτυξη και την προώθηση αυτού του ευρωπαϊκού παραδείγματος που είναι εκπαίδευση και κατάρτιση διαβίου που θέλει να είναι επικοδομητική εν ώψη της απασχολησιμότητας. Αυτό συνέβη για αρκετά χρόνια και φυσικά ε, είχε απομακρυνθεί πολύ από το αρχικό πνεύμα του συστήματος στην Γαλλία. Ε, είμαι ιδιαίτερα ε, διάκυμε μάλλον ιδιαίτερα θετικά πάνω για το ζήτημα για την ε, αξιολόγηση αυτής της ε, διαβίου μάθησης και της απασχολησιμότητας. Θα προσπαθήσω να σας το καταδείξω ότι εντάσσεται σε ένα σχολικό σύστημα το οποίο αν το δούμε από άλλη προπτική γωνία δείχνει ιδιαίτερα περίπλοκο αλλά αυτή η περιπλοκότητα αποτελεί και μια πηγή πλούτου για να βρούμε πόρους για την εξέβρεση διαφόρων εμπειριών προκειμένου να υπηρετήσουμε αυτή την ιδέα της διαβίου μάθησης. Το σύστημα δευτερεύουσας εκπαίδευσης στη Γαλλία είναι σχετικά περίπλοκο. Έχουμε έναν προσανατολισμό που ξεκινάει από την ηλικία των 15 ετών και οι νέοι οδηγούνται στο να εγγραφούν σε επαγγελματικό δίκτυο, ε, ε, ε, λύκειο ή σε ένα λύκειο το οποίο θα οδήγησε σε τεχνολογική ή γενική ε, κατάρτιση. Είναι ένα σύστημα λοιπόν κάπως περίπλοκο, μόνο ότι η τεχνική κατάρτιση θα οδηγησε σε τεχνολογικη η γενικη καταρτιση ειναι ενα συστημα λοιπον καπως περιπλοκο μόλις οτι η τεχνικη καταρτιση θα προσεγγισει την γενική προσέγγιση. Μετά έχουμε και ένα σύστημα περίπλοκο με το μπακαλωρεά για να μπορείς να μπει κάποιο παιδί στο πανεπιστήμιο και το, σε υπόλοιπε σχολές ε, που ονομάζουν, ονομάζουμε Grand École, μεγάλες σχολές, οι οποίες ε, συχνά ε, έχουν άμεση σχέση με την ιστορία της χώρας μου, ειδικά με την Γαλλική Επανάσταση, όπου ε, προκειτώ να εκπαιδευτούν τα νέα στελέχη μιας σύγχρονης χώρας. Θα καταλάβατε ότι από τώρα η προτεραιότητα αποδίδεται στα διπλώματα, κάτι το οποίο απομακρύνει την ε, πορεία ενός νέου και ε, δημιουργεί διάφορες εμπειρίες επαγγελματικέ ε, ή μη και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν από την ιδέα ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την διαβίου κατάρτιση, διαβίου μάθηση και την αξιοποίηση κάποιων πτυχών. Ο νόμος του 2013 ανέθεσε σε εμπειρογνώμονε την κατάρτιση μιας στρατηγικής ε, της εκπαίδευσης. Οι εργασίε ε, υποβλήθηκαν πριν από δύο μήνες ε, και θα πρέπει λοιπόν να αποσυνδεθεί η αρχική εκπαίδευση που οδηγεί στο δίπλωμα με την διαβίου μάθηση, με τη συνεχή μάθηση, κάτι το οποίο θα λάβει υπόψη τα κεκτημένα και της όλης εμπειρίας του προσώπου και η ενότατη εκπαίδευση θα πρέπει τα προσεγή χρόνια να αναπτύξει την εναλλαγή, δηλαδή μια εκπαίδευση η οποία γίνεται ανάμεσα στην αρχική εκπαίδευση ή την πανεπιστημιακή και αυτή που δημιουργείται στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που ονομάζεται στην Ευρώπη ε, ε, κατάρτιση διτή σας μίλησα τώρα για την ανώτερη εκπαίδευση. Επίσης αυτή η προσπάθεια πλούστευσε τα πανεπιστήμια δημιουργώντας ε, μεγάλους ε, πανεπιστημιακούς πόλους, ε, μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα. Έχουμε και επίσης περιοχές που παρέχουν υπηρεσίες προσανατολισμού. Παράλληλα σε αυτές τις υπηρεσίες υπάρχουν εδώ και 15 χρόνια αυτό που ονομάζουμε ΔΕΑ, ε, δηλαδή αξιοποίηση των ε, κεκτημένων της εμπειρίας που ανταποκρίνεται σε αυτή τη σύσταση του 2012 που είναι να αποκτήσει κάθε ευρωπαϊκό κράτος ένα σύστημα αξιολόγησης των ε, κεκτημένων της εμπειρίας και της κεκτημένης προκειμένου να αξιοποιήσουμε την εναλλαγή και όλα τα συστήματα κατάρτισης που ανέφεραν οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα με την προσφυγή στο ψηφιακό κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Φραντσέσκα Πουλιέζε έχει το λόγο από την γερουσία της Ιταλίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ιταλική κυβέρνηση μετά από πολλά έτη περικοπών αποφάσισε να επενδύσει σημαντικά στο ζήτημα της κατάρτισης διότι θεωρούμε πως η καλύτερη δομική πολιτική για την καταπολέμηση της, της ανεργίας των νέων και των κοινωνικού αποκλεισμού είναι η επένδυση στην εκπαίδευση. Ο, ο ο οργανισμός 107 που εγκρίθηκε από την Ιταλική Βουλή φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή και εφαρμόζεται από φέτος, από το φετινό σχολικό έτος, έχει ως στόχο την μείωση της εγκατάλειψης ε, στο σχολείο και την καλύτερη εκπαίδευση σε θέματα φυσικής και μαθηματικών, η βελτίωση στην εκπαίδευση πρώτη φάση σχολικής εκπαίδευσης, αυτό θα ξεκινήσει αργότερα, η βελτίωση της επαγγελματικότητας των καθηγητών, των εκπαιδευτών, να πω επίσης ότι ακούσαμε από τους ίδιους τους δασκάλους ε, ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία οδηγούν σε ανταλλαγές με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία είναι η καλύτερη εμπειρία για την ε, περαιτέρω κατάρτισή τους και αυτοί που αξιολογούν θετικότερα. Επίσης η βελτίωση των εγκάρσεων ικανοτήτων των παιδιών και η βελτίωση των δυνατοτήτων απασχολησιμότητας. Αυτό έγινε μέσω μιας ε, επένδυσης τριών δις ε, ευρώ μέσω της ε, πρόσληψης 40.000 καθηγητών και με την ε, εναλλαγή σχολείου ε, ε, χώρου εργασίας 400 ώρες για τα τεχνικά και τα κλιματικά διλίκια και 200 ώρες για τα λύκεια. Κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό ως δραστηριότητα όχι μόνο εκπαιδευτική αλλά και προσανατολισμού για τις περαιτέρω επιλογές των παιδιών αυτό είναι μια απόλυτη καινοτομία για το Ιταλικό σύστημα. Επίσης υπάρχει και κάτι ακόμα Μιλάω για το εθνικό πρόγραμμα για το ψηφιακό σχολείο. Το 90% των σχολείων ήταν συνδεδεμένο με το διαδίκτυο, αλλά μόνο το 7% των ε, σχολικών αιθουσών ήταν συνδεδεμένο με το δίκτυο. Τα υπόλοιπα ήταν ε, ε, αίθουσες ε, των καθηγητών κλπ. Η κυβέρνηση λοιπόν θα επενδύσει μέσα σε τέσσερα χρόνια και έτσι όλα τα σχολιά θα συνδεθούν με το δίκτυο έτσι ώστε η ψηφιοποίηση να αποτελέσει ένα κίνητρο για την καινοτομία, τη διδακτική καινοτομία. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να επενδύσουμε 40 εκατομμύρια ευρώ για την κατάρτιση των ε, καθηγητών και 90 εκατομμύρια ευρώ όχι μόνο για τη δημιουργία εργαστηρίων αλλά και για την ε, συμπερίληψη του ψηφιακού εκπαιδευτή σε κάθε σε κάθε ε, σχολείο. Κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό, το οποίο άκουσα και εδώ με πολύ ενδιαφέρον, για να βελτιωθούν οι εγκάσεις ε, δυνατότητες των παιδιών είναι η ενίσχυση της ε, προσφοράς ε, κατάρτισης για τους φοιτητές μας ξεκινώντας από την μουσική. Ακούσαμε πριν το έξοχο πρόγραμμα μουσική που διδάσκεται από εξειδικευμένους δασκάλους από το δημοτικό, την τέχνη, το αγγλικά, αλλά και εμπειρίες ε, σχετικά με την ενεργό ηθαγένεια ή την ε, ενεργό ιδιότητα πολίτη. Πρέπει να δημιουργήσουμε συνειδητούς πολίτες. Ε, αυτή η επένδυση απαιτεί μια συμμετοχή των σχολιών αλλά και μια λογοδοσία από πλευράς τους. Επίσης ε, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στο Ιταλικό σύστημα και ένα σύστημα αξιολόγησης, πρώτα απ' όλα αυτοαξιολόγησης των σχολείων, αξιολόγησης ε, των ε, διευθυντών των σχολείων ανά τριετία και αξιολόγηση των καθηγητών που θα λαμβάνουν και με ένα πριμ για την εργασία τους και για την αξία τους, κάτι το οποίο δεν είναι φύστατο στο Ιταλία και νομίζω ότι ήμασταν οι μοναδικοί στην Ευρώπη που είχαμε ως μοναδικό κριτήριο για την προαγωγή των, ε, των καθηγητών το κλιμάκιο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόσφατη η μεταρρύθμιση, αλλά ξεκίνησε με άμεση εφαρμογή από φέτος. Το λέω με υπερηφάνεια ως Ιταλία, διότι σε πολλά κράτη υπόθηκε ότι αυτές τις χρονιές κρίσης κάναμε περικοπές στην εκπαίδευση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στη χώρα μου το έπραξαν, όπως και άλλα κράτη, όπως η Ελλάδα για πολλά, πολλούς λόγους, όχι μόνο η Ελλάδα, όλα κράτη τα οποία θα μπορούσαν και να μην το πράξουν είδαμε ότι είχε καταστροφικές ζητώσεις και στο θέμα της ε, κοινωνικής ανισότητας. Αυτή λοιπόν η επανεπένδυση στην στην ε, επανεπένδυση στην κατάρτιση και την εκπαίδευση είναι κάτι το θετικότατο. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Τζέραρτ Κράουφουέλ, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά από την γερουσία της Ιρλανδίας. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σωστά προφέρατε το όνομά μου. Εγώ ασχολούμαι με τη διαβίου κατάρτιση όλη μου τη ζωή. Μου έδωσε την ευκαιρία να αλλάξω δουλειά 11 φορές και να καταλήξω τελικά μέλος της, ε, Ιρλανδία, της Ιρλανδικής Γερουσίας. Κοιτάξτε, η προσπάθεια της ε, τωρινής γενιάς ε, να εκπαιδευτεί στην Ιρλανδία ήταν πάρα πολύ επιτυχής. Ε, ο σάμας μας λέει πως γύρω στο 90% των παιδιών στην Ιρλανδία τελειώνουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ο μεσόρος του ΟΣΑ είναι 83%, επίσης 51% ε, πήγαιναν στην ε, ανώτατη εκπαίδευση. Το μέσο όρο του ΩΣΑ είναι 41%. Ξέρουμε πως όλες τις χώρες του ΩΣΑ οι ενήλικες με τριτοβάθμια εκπαίδευση κερδίζουν περισσότερα από τους ενήλικες με δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αυτοί με τη σειρά τους κερδίζουν περισσότερα με αυτούς που έχουν την ε, βασική εκπαίδευση. Οπότε εξακολουθούμε να θεωρούμε την εκπαίδευση ως επένδυση στο μέλλον και στην απασχόληση. Όμως η πολιτική δεν έχει μόνο οικονομικούς στόχους, ε, πέρα από την προσωπική και εθνική ευημερία υπάρχουν ευρύτεροι στόχοι να αυξηθεί το κοινωνικό κεφάλαιο, η ευημερία, η εμπιστοσύνη, η δημοκρατία και η κοινωνική συνοχή. Και πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ ακολουθούμε ε, τις γενικές τάσεις, πως ε, τα ποσά του πληθυσμού με τον υψηλότερο αλφαβητισμό και εκπαίδευση έχουν και τα υψηλότερα ποσοστά εθελοντισμού και προσωπικής εμπιστοσύνης κτλ. Αυτά είναι θετικά, αλλά παρόλα αυτά η ανεργία των νέων στην ε, Ιρλανδία είναι 19,5% είναι 8,5% για το σύνολο του πληθυσμού οπότε δεν πρέπει να και είχαμε σημαντικές βελτιώσεις παρόλα αυτά από το 2011 όταν η ανεργία των νέων ήταν 31% μιλάω ιδιαίτερα για τους νέους που δεν ε, ολοκληρώνουν την ε, δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή όταν τελειώνουν δεν προχωρούν στην τρίτο βάθμια. Η Ιρλανδική τριτο η ιρλανδικη κυβερνηση με διακομματική συνένεση ανταποκρίθηκε με το να συστήσει την αρχή για την διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι μέχρι το 2011 η εκπαίδευση και η κατάρτιση στο επίπεδο μετά δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν σε δύο υπουργεία η επαγγελματική κατάρτιση και που ήταν στο Υπουργείο Παιδείας, και το κομμάτι που ήταν ε, στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Πρόνοιας. Αυτά τώρα συγχωνεύτηκαν ως αρμοδιότητα και σκόπευα να μπω και σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το τι κάνει η αρχή ε, εκπαίδευση και κατάρτισης, αλλά θα με συγχωρέσετε τώρα γιατί άλλαξα λίγο κάποια από τα πράγματα που ήθελα να πω και ίσως ακουστεί περίεργη ομιλία μου. Κοίταξτε, είχαμε ένα πρόγραμμα μαθητείας το οποίο γίνεται και επιτόπου στους τόπους εργασίας και θεωρητικά μαθήματα και αφορούσε νέους οι οποίοι εγκατέλειπαν την επίσημη εκπαίδευση και στόχο έχουν να δοθεί κάποια κατάρτιση και κάποια εργασιακή εμπειρία. Παρόμοιο πράγμα στις ε, κοινότητες ε, το οποίο παρέχουν οι κοινότητες και όχι εκπαιδευτικοί και ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα που είχαμε ως αποτέλεσμα του Κράχα, ένα πρόγραμμα ονόματι Momentum το οποίο είναι σημαντικό γιατί πάνω από 50% των ε, συμμετεχόντων έχουν φύγει από το Ταμείο Ανεργίας. Βλέπουμε όμως πως τα προγράμματα αυτά πράγματι αφορούν αυτούς που ωφελούνται από αυτά. Και πρέπει να συνεχίσουμε και για τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Και μέχρι πέρσι ε, εγώ ήμουν στον τομέα της εκπαίδευσης και βεβαίως η χρηματοδότηση στην εκπαίδευση πηγαίνει με βάση την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων, αριθμός διδασκομένων, ε, πόσες εκπαιδευτικές μονάδες συγκέντρωσαν και τα λοιπά διπλώματα και, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Πράγματι ισχύει αυτό, αλλά κάπου ξεχνάμε την συγκεκριμένη ομάδα, γιατί είπα ότι 90% ολοκληρώνουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 10% που δεν ολοκληρώνει την ε, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μικρή αυτή ομάδα που ξεκίνησαν ε, να δουλεύουν ειδικά μετά το κράχ και που ε, έπιαναν καλοπληρωμένες ε, χειρονακτικές δουλειές έχουν πλέον χάσει την θέση τους στην αγορά εργασίας και σε μεγάλο βαθμό έχουν χάσει τις βασικές δεξιότητες που είχαν όταν έφυγαν από την εκπαίδευση. Οπότε τώρα βρίσκονται σε μια θέση όπου έχουν περιθωριοποιηθεί και οι εναλλακτικέ είναι είτε τα επιδόματα πρόνοιας είτε το έγκλημα. Μιλάμε για μικρό ποσοστό αλλά σημαντικό. Και ακούσαμε και για αυτά τα οποία έγιναν στην Γαλλία και οι περιφερειοποιημένοι κινδυνεύουν ε, να ριζοσφαστικοποιηθούν και αυτό πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Λοιπόν, η διαβίου κατάρτιση ε, σημαίνει πως ε, θα πρέπει να σημαίνει πως υπάρχουν οι βασικές δεξιότητες για να έχει κανείς πρόσβαση στο πρόγραμμα. Πολλά προγράμματα σβήνει το μικρόφωνο του ομιλητή. Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, για να μπει κανείς σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να υπάρχουν ε, οι βασικές δεξιότητες, ε, αλφαβητισμός, αριθμητική κτλ. Τα προγράμματα λοιπόν τα οποία έχουν ως στόχο μετρήσιμα αποτελέσματα δεν καλύπτουν αυτό την πτυχή. Τα κοιτάμε πολύ με μια λογιστική, αν θέλετε, σκοπιά. Πρέπει να αναπτύξουμε κάποια προγράμματα όπου το μόνο αποτέλεσμα θα είναι η ολοκλήρωση, χωρίς αξιολόγηση, απλά να τα ολοκληρώσει κανείς. Και αν θέλουμε να μετρήσουμε κάτι, θα μετράμε το πόσοι πήγαν μετά σε επίσημη εκπαίδευση, όπου υπάρχουν μετά επίσημα προσόντα και τίτλοι σπουδών. Ε, το βάρος λοιπόν που πρέπει να δοθεί, όπως ε, είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι να έχουμε σωστούς ενεργούς ε, πολίτες στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο. Δύο βουλευτές και ζητήστε λόγο και το Youth Forum αλλά 12 και 30 θα πρέπει να ξέρετε πως ε, δεν θα έχουμε πλέον διερμηνία. Είστε σύντομοι, λακωνικοί. Λάουρα Λόπες από το Youth Forum. Ευχαριστώ. Όταν ρωτήσαμε τους νέους με τους οποίους δουλεύουμε πού απέκτησαν τα καλύτερες δεξιότητές τους, η απάντηση σχεδόν πάντα είναι εκτός σχολείου. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, την εκπαιδευτική αξία των ε, ενώσεων νέων και δεύτερον ότι χρειάζονται αλλαγές στο σύστημα επίσημης εκπαίδευσης. Μην ξεχνάμε ότι η αποστολή της εκπαίδευσης επίσημης και άτυπης είναι να αναπτύσσει δεξιότητες για τη ζωή δηλαδή και για την προσωπική και για την επαγγελματική ζωή έτσι ώστε οι νέοι να έχουν αξίες και γνώσεις και δεξιότητες για να ζήσουν τη ζωή τους αξιόπρεπα, αξιοπρεπώς. Συγγνώμη. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ικανότητες και για να μάθουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας και για να μαθαίνουμε. Να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, αλλαγές και να μπορούμε να αρπάξουμε τις καινούριες μας ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει κατανόηση ότι έχουμε μια κοινή ευθύνη και με τους παρέχοντες ε, επίσημη και άτυπη εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης για τους νέους και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Νομίζω ότι ο νέος στόχος 4-7 ε, ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης είναι εξαιρετική ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν και αυτά ευθύνη, κοινή ευθύνη να εξασφαλίσουν αυτό το πράγμα και σε εθνικό επίπεδο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση του συνόλου της. Ε. Ευχαριστώ και τώρα δύο ακόμα παρεμβαίνοντες. Σβέρ, συγγνώμη, Γιάννη Μάντισον από την Εστονία και μετά ο δικό μου συνάδελφος. Ε, ευχαριστώ. Για να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση, εμείς στην Εστονία πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μαθαίνουμε ένας από τον άλλο, ιδιαίτερα από ε, ιδιαίτερα ε, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης το πρόβλημα είναι πιο σημαντικό, πιο οξύ. Εμείς στην Εστονία έχουμε ένα σύστημα συνεργασίας ανάμεσα στους εργοδότες και τα συστήματα κατάρτισης και επιμόρφωσης. Γιατί όταν μιλάμε για μαθητεία και στάζ ε, θα πρέπει να δίνουμε στους ε, σπουδαστές ε, ευκαιρίες να εργαστούν σε επιχειρήσεις. Αυτό θα κάνουμε τα επόμενα τρία χρόνια στην Εστονία. Θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίες να εργαστούν σε επιχειρήσεις μέσω συνεργασιών. Θα πρέπει να δώσουμε τέτοιες ευκαιρίες ιδιαίτερα και στους ανθρώπους που έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, έχουν πάρει ένα τίτλο, ένα πτυχίο, αλλά δεν έχουν ακόμα αποκτήσει εργασιακή εμπειρία. Θα πρέπει και σε αυτούς να δώσουμε ευκαιρίες και βέβαια σε αυτούς που ακόμα σπουδάζουν. Ο, ο Γάλλος βουλευτής Yves έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να εκπαιδεύει τους νέους σε, σε επαγγέλματα τα οποία δεν ε, υπάρχουν καν τώρα. Θα πρέπει να να αρχίσουν να προσαρμόζονται στις εργατικές ε, στις ανάγκες εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν το ψηφιακός Χαρακτήρα θα πρέπει να είναι, μπορεί μάλλον να είναι ένα, ένα διαπαιδαγωγικό εργαλείο σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ με τρόπο προοδευτικό και αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στον τελευταίο μιλητή που μίλησε για τους ε, μαθητές. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα οργάνωσα ένα συνέδριο με κάποιες επιχειρήσεις και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Όπως ξέρετε στην Ευρώπη υπάρχει ήδη μια συμμαχία για τους ε, μαθητές από το 2013 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολλές επιχειρήσεις συμμετέχουν ε, και δίνουν στους νέους ε, δουλειά και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες νέους. Έτσι οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες ε, που τους χρησιμεύουν στην αγορά εργασίας. Έτσι μπορούμε να διευκολύνουμε τη μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας. Και θεωρώ πως αυτό είναι σημαντικό και για τις προκλήσεις ε, του μέλλοντος. Επίσης, ε, τα αισθήματα του σχολείου θα δώσουν τους νέους, στους νέους την ευκαιρία και να ενταχθούν. Ευχαριστώ κυρία Σοντρόβα. Πολύ σύντομα παρακαλώ γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα φύγουν οι Ευχαριστώ για τις ψηφοφορίες ε, που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Να προσθέσω όμως, γιατί όλοι μιλούσατε για γνώσεις, ε, νέες ικανότητες, εκπαίδευση των ε, δασκάλων στη Γαλλία, αλλά υπάρχουν νέες ανάγκες για τα σχολιά, αλλά και για να εργαστούμε πάνω στα θέματα της άτυπης εκπαίδευσης απαιτείται να χρησιμοποιήσουμε στο σχολείο και τα αποτελέσματα της τυπικής εκπαίδευσης. Η εξαίρεση της Φιλανδίας Γνωρίζω ότι σε εσά η μισθή των καθηγητών είναι υψηλότερη των υπολείπων. Αλλά στα άλλα κράτη γνωρίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με τους μισθούς των καθηγητών και των δασκάλων. Εσείς είστε ικανοποιημένοι με τις αμοιβέ. Πρόεδρος, παρακαλώ να είστε λακωνικοί. Ένα λεπτό, όχι παραπάνω, λοιπόν, διαφορετικά σας διακόπτω. Ευχαριστώ. Κύριο Στάρκουλα. Τρεις ερωτήσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την εσωτερική αγορά της οποίας αρχή είναι η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Οπότε εμείς εκπαιδεύουμε το εργατικό δυναμικό για όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Και η εκπαίδευση αυτή τη στιγμή αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ήπια ε, ισχύ, ε, δηλαδή συντονισμό κατά βάση των εθνικών πολιτικών. Οπότε η ερώτησή μου είναι εξής. Ποια είναι η γνώμη σας, χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή ακόμα και νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπαίδευση και αν ναι, τι είδου συνεργασία χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Thanks. Thank you. Ε, Julie. Julie. Συγγνώμη που βιάστηκα προηγουμένω, Είναι πολύ ωραίο που ακούμε νέου ανθρώπους εδώ για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Νέους και οργανώσεις νεολαίων. Οι... Αυτές οι οργανώσεις τις τελευταίες δύο μέρες διοργάνωσαν διάφορες εκδηλώσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε θέλω να, πω, να ρωτήσω το εξής. Ε, ε μάλλον να ζητήσω από τους πολιτικούς σε όλα τα επίπεδα να ακούν τους νέους γιατί εμείς έχουμε πιο πολλά να μάθουμε από αυτούς από ό,τι αυτοί από εμά. Και ποτέ δεν έχουμε σεβαστεί αρκετά ε, τις δεξιότητες, ικανότητες ε, και την επιμονή που φέρνουν αυτές οι οργανώσεις νέων. Δεύτερον, ε, δημιουργικότητα και τέχνη. Ε, δεν είπαμε αρκετά για αυτό το θέμα. Είναι εργαλεία τα οποία είναι ε, δυνατόν να μεταφερθούν και να κινηθούν μέσα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε βοηθούν στην ε, απασχολησιμότητα. Και ε, νομίζω θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση για τον δια, διαπολιτισμικό διάλογο. Τώρα αν υπάρχουν απαντήσεις ε, σε ελάχιστα λεπτά. μόνο αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Διαφορετικά δεν χρειάζεται να λάβετε το λόγο, διότι θα πρέπει να δώσω το λόγο στον κλείνω μικρόφωνο Πρόεδρο, στον κύριο Χάρα Γκρούμπερ, είναι πολύ... πρόκειται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επικεφαλής της ψηφιακής οικονομίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, θα σα δώσω το λόγο, αλλά πρέπει να απαντήσουν. Okay, I changed place. Thank you very much your place. Uh, uh, uh, about digital schools. I think so that's the future. And, uh... Μιλήσαμε για τα ψηφιακά σχολεία και πραγματικά πρέπει να αποκτήσουν ε, ε, δυνατότητες οι δάσκαλοι. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας στη Φιλανδία τα επόμενα χρόνια. Πώς θα αλλάξουμε την ε, εκπαίδευση των καθηγητών και τι ικανότητες χρειάζονται. Κάτι το οποίο δεν έχουμε συζητήσει εδώ πέρα αφορά την εκπαίδευση των συνταξιούχων. Γιατί υπάρχουν συνταξιούχοι που θέλουν να απασχοληθούν και θα πρέπει να έχουν και αυτοί τις ε, δυνατότητες να μάθουν νέες δεξιότητες και να μπουν στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ για την απάντηση. Άλλος, κλείνει το μικρόφωνο του Προέδρος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το μικρόφωνο μου. Οι διερμηνείς μπορούν να παραμείνουν πέντε λεπτά ακόμα, αλλά και μετά θα συνεχίσουμε στα αγγλικά. Στο τέλος έχουμε να βγάλουμε για την οικογενική φωτογραφία, μην το ξεχνάμε. Πέραν του ότι πρέπει να γευματίσουμε. Ξέρετε πως ε, υπάρχει αυτό το έκτακτο πρόγραμμα επενδύσεων στην Ευρώπη που ανέρχεται σε 24 δις προς το παρόν. Αλλά ελπίζουμε να μπορέσει να προκαλέσει μέσω συγχρηματοδοτήσεων με τον ιδιωτικό τομέα να φτάσει λοιπόν γύρω στα 300 δις προγράμματα που θα έχει προετοιμάσει η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο όρος education. Εμείς θα πρέπει να το προσέξουμε και να το προασπιστούμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα διακυβέρνησης τόσο ανάμεσα σε εθνικά κοινοβούλια αλλά και σε εθνικές κυβερνήσεις όπως είπε ο κ. Ντουράν και άλλοι για να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο διότι υπάρχουν κάποιες στρατηγικές που θα πρέπει να υλοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες δίνοντας βεβαιότητα και στους ιδιώτες επενδυτές ότι η Ευρώπη θέλει να ακολουθήσει αυτήν την οδό και να δεχθεί αυτό το έκτακτο πρόγραμμα επενδύσεων συμπληρωματικό του πολιετούς προγράμματος ως ένα ποιοτικό άλμα και να καλύψει τα κενά, τα χάσματα που υπάρχουν. Το ένα αυτό, ένα αυτά είναι το ε, ευρυζωνικό ζήτημα το ψηφιακό και μπορεί και ο Γκρούμπερ να μας πει το τι πράττει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και εμείς ε, θα θέλαμε να συνεχιστεί ή να υπάρξει συνεργασία και με τα Ευρωκοινοβούλια όπως και με τα εθνικά. Ευχαριστώ. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας ε, μιλήσω. Λοιπόν, σύντομα θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά τα θέματα. Η τράπεζα μας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ιδιοκτησία δηλαδή των κρατών μελών και χρηματοδοτεί έργα. Και για να είναι ένα έργο επιλέξιμο πρέπει να είναι επιλέξιμο πρώτα απ' όλα ως ε, πολιτικός στόχος, θα σας πω σε λίγο γι' αυτό, αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι οικονομικά, τεχνικά και δημοσιονομικά βιώσιμο. Αλλιώς δεν μπορεί η τράπεζα να χρηματοδοτήσει. Λοιπόν, όσον αφορά τα ποσά, το τι χρηματοδοτεί μάλλον η τράπεζα στον τομέα της εκπαίδευσης βλέπετε πως είναι κυρίως υποδομές γιατί αυτό περισσότερο ταιριάζει σε μακροπρόθεσμα δάνεια και το σημαντικό είναι πως η Ευρώπη δεν επενδύει αρκετά στις υποδομές για την εκπαίδευση. Κατά κανόνα είναι 10% του προπολογισμού της ε, εκπαίδευσης, αλλά de facto τα τελευταία χρόνια έχουμε υπολογίσει πως υπάρχει... Δεν, υπάρχει αρκετή... Ε, δεν υπάρχουν αρκετές δαπάνες σε αυτό το τομέα και απαιτούνται να αυξηθούν για τις υποδομές μιλάμε, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν γίνεται σωστή εκπαίδευση σε ακατάλληλη υποδομή. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τι έχει κάνει η τράπεζα τα τελευταία χρόνια, γύρω στα 5 δισεκατομμύρια στον τομέα της εκπαίδευσης, ε, ειδικότερα στις υποδομές και βλέπουμε επίσης τον δανεισμό στον ε, τομέα αυτών και βλέπουμε πως ε, αυξάνεται και θα συνεχίσει να αυξάνεται γιατί υπάρχει σοβαρή ανάγκη για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ε, οπότε εξοδεύουμε σε υποδομές που ουσιαστικά είναι μια επένδυση για το μέλλον και αποδεδειγμένα επιδρούν στην οικονομική ανάπτυξη. Τώρα, να πω λίγα πράγματα για μια νέα πρωτοβουλία που ανέλαβε η τράπεζα για τις ε, θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες, συγκεκριμένα για το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Το είδαμε από δύο πλευρές. Το ένα είναι η πλευρά της ζήτησης ε, και το άλλο της προσφοράς. Το ζήτημα λοιπόν τη ζήτηση είναι το ποιο απασχολεί του νέου ε, κυρίω οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν κατά κύριο λόγο τους ε, νέου και είναι και πιο ευέλικτε. Και στην πλευρά της ε, προσφοράς βλέπουμε το τι κάνουν, τι μπορούμε να δώσουμε στην αγορά εργασίας. Πρέπει οι νέοι να έχουν δεξιότητες που είναι χρήσιμες στην αγορά εργασίας. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο πυλώνες επί των οποίων ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία με την ε, Κομισιόν αρχικά με 6 δισεκατομμύρια από την Κομισιόν και άλλα τόσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η επένδυση λοιπόν αυτή είχε στόχο κυρίως τις υποδομές, τις εκπαίδευση και πρωτοβουλίες που θα δώσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την αγορά εργασίας. Βλέπουμε εδώ πέρα τα περισσότερα πράγματα. Οπότε δίνουμε και δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό τον όρο ότι θα προλάβουν νέους ή θα παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τα υπόλοιπα ε, βλέπετε πως είναι γύρω στα 3 δισεκατομμύρια το έτος. Η συζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε, οπότε ήταν πολύ επιτυχημένο το πρόγραμμα. Και έγινε και μια μελέτη ανεξαρτήτων συμβούλων που μπορώ να σας την ε, δώσω εάν ε, ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας για την νεολαία. Αυτά θα σταματήσω εδώ. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σημαντικά όσα μας είπατε. Η σας ευχαριστεί τους Γερμινείς και οι Γερμινείς ευχαριστούν την πρόεδρο. Δυστυχώς πρέπει να σας αφήσουμε. Θα συνεχίσουμε στα αγγλικά. Very interesting to know uh, just one thing if you have just one minute or I imagine that you are, you are interested like me just to know how uh, we